Συνεχίζουμε λοιπόν από τα χθε και είμαστε τώρα στο σημείο της ημέρα της διάταξης υπαριθμών 19. Η πρώτη συζήτηση για μια νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με την πιστοποίηση των ορυκτών που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και που συνδέονται με υψηλό κίνδυνο να έχουν εξοριχθεί σε συνθήκες σύγκρουσης και αναφερόμαστε κυρίως ε, για τα ορυκτά από τη Δημοκρατία του Κονγκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι πρώτες ύλες μας δεν ε, αποκτώνται με τρόπους οι οποίοι είναι απαξιωτικοί για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε ζώνες πολέμου. Είναι πολύ <clears throat> καλό λοιπόν το ότι έχουμε μία πρόταση νομοθετική από την πλευρά της Κομισιόν. Και υπάρχουν αντίστοιχες ε, ρυθμίσεις σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως ο νόμος Dodd-Frank στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και έχουμε φυσικά και τον εισηγητή μας, τον κύριο Βίνκλα, αλλά είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μπορεί, θα μπορούσε να μας παρουσιάσει εν συντομία και πάλι την πρότασή της, ο κύριος Πέτρος Σουμίλης. Yes, good morning. Uh, Καλημέρα σας. Με μεγάλη χαρά κάνουμε εδώ την πρώτη συζήτηση στην Επιτροπή σας για το σχέδιο κανονισμού που υποβάλαμε σχετικά με την υπεύθυνη εισαγωγή ορισμένων μετάλλων του ξτενίου, ταντάλου και άλλων και χρυσού. Όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε, Το έχουμε υποβάλει και το έχει συζητήσει το Κοινοβούλιο. Υπήρξαν αρκετά ψηφίσματα. Είναι πρόταση που την προετοιμάσαμε με μεγάλη προσοχή. Έγινε δημόσια διαβούλευση με πολλούς ενδιαφερόμενους και φυσικά κάναμε και μια πρώτη αξιολόγηση και μετά καταθέσαμε την πρότασή μας είναι πρόταση που βασίζεται στις διεθνείς προσπάθειες που προϋπήρχαν από άλλες διεθνείς οργανώσεις όπως τον ΟΣΑ και τον ΟΙΕ και προσπάθειες και από ορισμένε χώρες στις Ηνωμένε Πολιτείες όπως το νομοσχέδιο ΦΡΑΝΚ και ιδιαίτερα ψηφίσματα και οργανώσεις γύρω από τις μεγάλες λίμνες. Βασιστήκαμε λοιπόν σε αυτές τις προσπάθειες και ιδιαίτερα στις κατευθυντήρες γραμμές του ΣΑ για αυτά τα τέσσερα ορυκτά Πρέπει όμως ήδη να πούμε από την αρχή ότι παρά τις διεθνείς αυτές προσπάθειες και την αναδιόμενη διεθνή συνένεση δεν υπάρχει καμία δεσμε, κανένας δεσμευτικός διεθνής κανόνας. Αντίθετα από άλλα θέματα και το τομείς όπου υπάρχει ενωσιακή νομοθεσία για την προμήθεια ορισμένων υλικών όπως την ξυλία και συμπληρώνει το, η πρόταση αυτή όχι μόνο αυτές τις διεθνείς προσπάθειες αλλά και τις προσπάθειες που έγιναν και από ορισμένε επιχειρήσεις ήδη έχουν αναλυφθεί προγράμματα από μερικές εταιρείες όπως ίσως γνωρίζετε. Η νομοθεσία αυτή έχει τρεις στόχους συμπληρωματικούς ο ένας με τον άλλον και συνδεόμενους. Πρώτον, να σπάσει η σύνδεση μεταξύ της εξόριξης αυτών των μετάλλων και της χρηματοδότησης ορισμένων σειράξεων και συγκρούσεων ή επαπειλουμένων συγκρούσεων. Δεύτερος στόχος, να δημιουργηθεί μια αγορά στην Ένωση για υπεύθυνη εμπορία τέτοιων ορυκτών και τρίτον να βελτιωθεί η δυνατότητα της Ένωσης και των επιχειρηματιών της για την εφαρμογή άλλων πλαισίων due diligence όπως λέμε. Ανάλογες προσπάθειες με την νομοθεσία Dort Frank στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια δεν είναι απομονωμένη αυτή η νομοθεσία. Είναι ολόκληρη δέσμη και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία ιδιαίτερα αναφέρεται σε ορισμένα κίνητρα που χορηγούνται για να συμπληρωθεί η νομοθεσία αυτή και από άλλα μέτρα για να διευκολυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος πιστοποιήσεων που προτείνουμε εκεί μέσα. Το σχέδιο κανονισμού αναπροϊόν αναφέρεται σε αυτά τα τέσσερα ορυκτά που σας ανέφερα για τα οποία υπάρχουν κατευθυντήρες γραμμές του ΩΣΑ. Γεωγραφικός το σχέδιο κανονισμού έχει πολύ ευρία κάλυψη και σχετίζεται με όλες τις περιοχές όπου σημειώνονται συγκρούσεις ή επαπειλούνται τι αυτές και αναφέρει και συγκεκριμένες περιοχές το κείμενο. Αντίθετα με την νομοθεσία Dot Frank που αφορά μόνο την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Εδώ λοιπόν επιλέξαμε τη γραμμή, το πρότυπο του ΣΑ. Ευρία κάλυψη δηλαδή. Τώρα για το πεδίο εφαρμογής και το θέμα της αλυσίδας προμήθειών που στοχεύει η νομοθεσία μας θελήσαμε να στοχεύσουμε την μέση οδό των προμηθειών και μεταποιητών. Αυτό είναι το κλειδί, είναι το επίπεδο όπου μας λείπει μας λείπουν οι πληροφορίες και κάναμε συγκεκριμένη προσπάθεια αυτό το επίπεδο να στοχεύσουμε ιδιαίτερα ώστε να βελτιώσουμε έτσι και τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών ώστε να διατεθούν αυτές σε ολόκληρη την αλυσίδα. Και αυτό διαφέρει από το νομοθέτημα των Ηνωμένων Πολιτειών Dodd Frank Και σημαίνει ότι αφού στοχεύουμε αυτό το μέσο επίπεδο της αλυσίδας, η νομοθεσία αφορά πολύ λιγότερους μεταποιητές γιατί αυτά τα τέσσερα ορυκτά αντιπροσωπεύουν έως ε, επιχειρήσεις περίπου 4.500. Ο μηχανισμός που προβλέπουμε είναι αρκετά ευρύς, δηλαδή η εισαγωγή των τεσσάρων αυτών ορυκτών στην Ένωση μπορούν εθελοντικά αν θέλουν να, αυτοπιστοποιηθούν ως υπεύθυνοι εισαγωγή των προϊόντων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τις αρχές της due diligence ώστε τα αγαθά που αγοράζουν να πιστοποιούν ταυτόχρονα την προέλευσή τους αν προέρχονται ή όχι από περιοχές συγκρούσεων ή επαπειλουμένων τιούτων ώστε δηλαδή τα ορυκτά που αγοράζουν να είναι πιστοποιημένα καθαρά Όλα αυτά βέβαια δεν βασίζονται μόνο σε δηλώσεις των υπευθύνων αυτών εισαγωγέων, αλλά θα ελεγχθούν, ελεγχθούν από τις αρχές που στις διάφορες χώρες μέλη θα αναλάβουν την εφαρμογή του κανονισμού αυτού. Και φυσικά θα γίνουν και επιτόπιοι θα τα ελέγχουν οι ίδιοι εισαγωγεί, αλλά θα γίνουν και εξωτερικοί. Και αν δεν διαπιστωθεί ότι δεν είναι σωστή η πιστοποίηση τότε μπορεί να αφαιρεθεί αυτή. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν όσο το δυνατόν υψηλότερου επίπεδου πληροφορίες σας είπα ότι αφορά τους εισαγωγείς 400 άτομα περίπου δηλαδή και θέλουμε όσο δυνατόν περισσότεροι από αυτούς να εφαρμόσουν αυτήν την αυτοπιστοποίηση. Γι' αυτό δώσαμε και μερικά κίνητρα που εξηγούνται και στο κείμενο και στη δήλωσή μας. Ένας, ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι σε αιτήσια βάση θα δημοσιεύουμε τον κατάλογο των ε, εκείνων που εισάγουν μέταλλα προσλιώσιμο εφόσον βέβαια αποδειχθεί ότι προέρχονται από καθαρές περιοχές. Αυτό νομίζω θα πιέσει τους εισαγωγείς να εισάγουν από καθαρές περιοχές και τις άλλες εταιρείες να αγοράζουν από αυτούς τους καθαρούς εισαγωγείς και μεταποιητάς. Επίσης θα υπάρχουν κίνητρα με τη μορφή βοηθείας, στήριξης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν πιο εύκολα να κάνουν τους ελέγχους στα πλαίσια πάντα του προγράμματος Due Diligence. και η δήλωση που συνοδεύει τον κανονισμό μιλάει και για κίνητρα ως προς τις δημόσιες προμήθειες, ιδιαίτερα για την αγορά προϊόντων μεταποιημένων από δημόσιες αρχές μέσω της δυνατότητας να συμπεριλαμβάνονται ρήτρες ποιότητας των εισαγωγέων ή των εισαγωγών ώστε να διασφαλίζεται η αγορά υλικού που, έχει, που θα έχει ελεγχθεί με τα μέτρα due diligence. Η Κομισιόν δήλωσε ότι σκοπεύει να αρχίσει την εισαγωγή τέτοιων ρητρών και στα δικά της συμβόλαια δημόσιων προμηθειών. Και ζητάει και από τα άλλα όργανα αλλά κυριότερα από τις χώρες μέλη να συμπεριλάβουν τέτοιες ρήτρες στα συμβόλαιά τους. Τέλος, όλα αυτά δεν πρόκειται να λειτουργήσουν παρά εάν και επιτοπίως οι αρχές των χωρών μελών και οι αρχές των ε, περιοχών ε, όπου σημειώνονται συγκρούσεις και σειράξεις εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα για να γίνει πιο αποτελεσματική η λειτουργία και των δικών τους πιστοποιητικών συστημάτων γνωρίζουμε ότι πρόκειται για χώρες με πολύ μεγάλα προβλήματα και αστάθειες και ότι επομένως είναι βασικό το σύστημα να είναι ισορροπημένο, προοδευτικό και αρκετά ευέλικτο ώστε να μην διαταράξει περαιτέρω την ήδη δύσκολη κατάσταση που σημειώνεται στις χώρες αυτές εάν επέβαλε παραδείγματος χάρη πολύ μεγάλο βάρος στις τοπικές αρχές που ήδη δεν έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και με αυτά κύριε Πρόεδρε καταλήγω την παρουσίασή μου και αν έχετε απορίες με τα χαράς να σας τις λύσω. Ευχαριστώ και ο κύριος Βίνκλερ έχει τώρα το λόγο εισηγητής μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα και σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσίαση αυτής της πρότασης που έχουν εκπονήσει και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου με βοηθήσατε να αρχίσω την εργασία μου με αυτή την πρόταση. Τώρα, για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας απασχολεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους ε, εισαγωγείς σε παγκόσμιο επίπεδο ορυκτών τα οποία είναι γνωστά ως TNTG ψευδάργυρο, σταντάλιο, βολφράμιο, 20% του παγκόσμιου εμπορίου και 15% στα συγκεκριμένα αυτά μέταλλα και 15% του χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο <clears throat> βρίσκεται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε γι' αυτό το λόγο μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι παράγονται με υπεύθυνο τρόπο αυτά τα ορυκτά και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποια διαφωνία αν πω ότι ο στόχος αυτού του κανονισμού είναι να σπάσουμε τη σύνδεση μεταξύ της εξόριξης και της εμπορίας αυτών των ορυκτών και την όλη αλυσίδα χρήστης και τη χρηματοδότηση των ενόπλων συγκρούσεων. Το να σπάσουμε αυτό το, αυτή τη σύνδεση δεν είναι εύκολο, το καταλάβατε και από αυτά που είπε η Κομισιόν, αλλά Έχουμε εκθέσεις που καταδεικνύουν ότι κάποιος συνδυασμός μεταξύ εκμετάλλευσης φυσικών ε, πόρων και συγκρούσεων ισχύει για το 1 πέμπτο περίπου όλων των χωρών στον κόσμο. Είναι πολύ σοβαρό λοιπόν το πρόβλημα και θα πρέπει να βρούμε από την πλευρά της Επιτροπής μας μια λύση, δηλαδή μια υπεύθυνη προσέγγιση. Θα πρέπει να βρούμε μια βιώσιμη, εξισορροπημένη λύση σε σχέση με τον τρόπο που μπορούμε να δράσουμε για να έχουμε υπεύθυνη προμήθεια ορυκτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι και μερικά χρόνια μετά την οικονομική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι τρωτή σε ορισμένου οικονομικού τομεί και θα πρέπει να αναλύσουμε και αυτέ τι ε, δυσκολίε που προκύπτουν από τον τρωτό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει από την Κομισιό να αναλάβει δράση για το θέμα αυτό. Εξέδωσε ένα ψήφισμα για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές ε, εμπόλεμες και έχουμε τώρα ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο συνδυάζεται με μια κοινή ανακοίνωση η οποία ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα μιας δημόσιας διαβούλευσης που οργανώθηκε πέρσι. Πιστεύω ότι αυτή η πρωτοβουλία θα πρέπει να συναρμοστεί με άλλες πρωτοβουλίες και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραγματικά χάρη πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλε. Και η νομοθεσία θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι τα τωρινά συστήματα τα οποία βασίζονται στα διεθνή πρότυπα, παραγματικά το σύστημα ε, απαραίτητης ε, εποπτείας και ελέγχου του ΟΣΑ, ε, είναι συστήματα τα οποία έχουν ήδη παγκόσμια εμβέλεια. Ο κανονισμός ο οποίος προτείνεται είναι μια νομοθετική πράξη η οποία θα είναι άμεσα εφαρμοστή στα κράτη-μέλη και η απόψή μου σχετικά είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια σειρά διευκρίνησεων σε συγκεκριμένα σημεία. Για παράδειγμα, θα αποτιμούσαμε να σαφή ορισμό για το ποιες είναι οι περιοχές οι οποίε πλήττονται από συγκρούσεις και υπέχουν υψηλό κίνδυνο. Επομένως θα πρέπει να καθορίσουμε σαφώς ποιο είναι το γεωγραφικό πλαίσιο, η γεωγραφική εμβέλεια αυτής της ε, νομοθεσίας. Και στη συνέχεια θα πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίζει ότι μια περιοχή είναι αντικείμενο συγκρούσεων και μετά θα πρέπει να έχουμε ως Κοινοβούλιο ε, κάποια διαβεβαίωση για τον κατάλογο των υπευθύνων χιτηρίων και κέντρων εξευγενισμού των μετάλλων. Να ξέρουμε πώς θα εκδίδεται αυτός ο κατάλογος, πώς θα ενημερώνεται, ώστε να μπορούμε να δώσουμε πράγματι τη διαβεβαίωση στις εταιρείε ότι θα έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν και να συμμορφωθούν με την νομοθεσία. Ο ορισμός του εισαγωγή επίσης είναι ο ακρογωνίος λίθος αυτού του νομοθετήματος και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε και εκεί πιο σαφείς. Και η αποτελεσματικότητα αυτού του κανονισμού θα προκύψει μονάχα αν έχουμε ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη και εάν ξέρουμε ποιος θα είναι και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην μελλοντική διαδικασία μετά την έγκριση αυτής της οδηγίας. Αναφέρθηκε και ο πρόεδρος και η Επιτροπή μας στην νομοθεσία George Frank στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία φυσικά επηρεάζει και τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να αναλύσουμε τα διάφορα μηνύματα τα οποία προέρχονται από τις ΗΠΑ που μας λένε ότι de facto ο νόμος Dodd Frank οδηγεί σε μια κατάσταση de facto εμπάργο στην γεωγραφική περιοχή των μεγάλων αφρικανικών λιμνών. Θέλουμε λοιπόν αυτό το εμπάργο ή πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό το οποίο είπε η Κομισιόν ότι ένας από τους στόχους και για μένα πιο σημαντικός στόχος αυτής της νομοθεσίας είναι να υπάρξει μια ευρωπαϊκή αγορά για ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων, τα οποία όμως την χάνουν υπεύθυνη εμπορία. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική μας για να παρέμβουμε και να βοηθήσουμε τις περιοχές αυτές και τις τοπικές κοινότητες να έχουν οικονομική βιωσιμότητα και να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη για την κοινή ανακοίνωση τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να υπάρξει αυτή η κοινή ανακοίνωση ταυτόχρονα με την πρόταση για τον κανονισμό. Η Επιτροπή μας λοιπόν θα πρέπει να έχει πάντα στο μυαλό της ότι εμείς συζητούμε ένα προτινόμενο κανονισμό. Φυσικά βέβαια θα πρέπει να κατανοούμε το ευρύτερο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μέτρα και τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, και οι δυνατότητες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικές. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην εξέταση αυτών των μέτρων και των κινήτρων που θα παρασχεθούν, γιατί ο στόχος μας είναι και πάλι να ενθαρρύνουμε το νόμιμο εμπόριο των ορυκτών αυτών, αλλά <clears throat> για παράδειγμα, σε σχέση με τα θέματα δημοσίων προμηθειών, που έχει πρόσφατα εξυγχρονίσει το πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρισκόμαστε σε μία φάση που τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτό το εξυγχρονισμένο πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχει νόημα να παρέμβουμε και πάλι στην εφαρμογή αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες ε, προμήθειες. Κλείνω λοιπόν κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας εάν με έχετε παρακολουθήσει, αλλά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα θα ήθελα να πω εν κατακλείδη ότι αποφασίσαμε να οργανώσουμε στην συνεδρία μας στις 3 και 4 Δεκεμβρίου μία δημόσια ακρόαση για το θέμα αυτό και ελπίζω θα προέλθει μεγαλύτερη σαφήνεια για το ζήτημα αυτό και θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Θα είναι παρόντες διάφοροι εμπλεκόμενοι και θα υπάρξει και η συζήτηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων με μέσα στην Επιτροπή μας για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης. Ευχαριστώ λοιπόν τέλος τον εισηγητή για την ε, της Επιτροπής ΔΕΒΕ για τα θέματα αυτά που είναι παρόν εδώ σήμερα και ελπίζω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία με αυτή την Επιτροπή στην προετοιμασία αυτού του φακέλου. <clears throat> Σας ευχαριστώ κύριε Βίνκλερ. Νομίζω ότι έχετε θίξει τα κύρια και κέρια σημεία αυτής της πρότασης και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε εντελεχώς την πρόταση της Κομισιόν. Χαίρομαι επίση για το γεγονός ότι μπορούμε να συνεργαστούμε στενά με την Επιτροπή ΔΕΒΕ για να δούμε και το θέμα της ανακοίνωσης και χαίρομαι που ο εισηγητής της Επιτροπής ΔΕΒΕ είναι παρόν ο κ. Βέντας, τον οποίο θα δώσω και το λόγο. Θέλω να σας ευχαριστήσω και αν μου επιτρέπετε θα χρησιμοποιήσω τα πολωνικά που είναι η μητρική μου γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι εισηγητής για την Επιτροπή ΙΤΕΒΕ. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Όπως βλέπουμε εμείς τα πράγματα, το θέμα των ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας τη Δευτέρα. Τώρα που σας μιλάω εκφράζω προσωπικές απόψεις αποκλειστικά. Οι αναπτυσσόμενες χώρες επειδή είναι συνήθως προμηθεύτες χώρες των ορυκτών αυτών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ε, τανταλίου ψευδαργύρου κλπ για σύγχρονες συσκευές Αυτές οι χώρες έχουν προβλήματα συγκρούσεων επίσης και πρέπει να δώσουμε σαν διεθνής κοινότητα μια απάντηση στο πρόβλημα. Είναι σημαντικότατο η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τη διεθνής νομοθεσία. Εμείς στην Επιτροπή μας προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να παρακολουθούμε την όλη αλυσίδα του εφοδιασμού για τα ορυκτά αυτά, από τη χώρα προέλευσης μέχρι την ε, Ευρώπη. Ο ρόλος του κυρίου Βίνκλερ εδώ είναι πολύ καλός, θέλω να το τονίσω, ο κύριος Βίνκλερ θέλει να σταματήσει ο εφοδιασμός ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων Ετοιμάζουμε γνωμοδότηση σχετικά με αυτό στην Επιτροπή μας. Αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι να συνεργαστούμε ε, σωστά γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Äh, Ευχαριστώ πολύ <clears throat> και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς έχουμε κάθε διάθεση να συνεργαστούμε με την Επιτροπή ΔΕΒΕ για να φέρουμε το πλοίο σε, στο σωστό λιμένα. Έχουμε 12 τώρα ομιλητές οι θέλουν να λάβουν το λόγο. 13. Προσφέρει κάτι περισσότερο. 14. 15. Τίποτα άλλο. Κάποιος άλλος θέλει να προσθεθεί. Και έχουμε άλλο ένα σημείο μέχρι την ψηφοφορία. Σας παρακαλώ λοιπόν να είσαστε σύντομοι. Δεν πρόκειται να σας περιορίσω. Αλλά άμα δείτε ότι προχωράει πάρα πολύ στο χρόνο η συζήτηση, θα πρέπει να είμαι πιο άκαμπτος. Η κυρία Κέτα από τους, η Αρένα, από τους ε, σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις που ακούστηκαν σχετικά με το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι σημαντικότατο ζήτημα. Αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάποια μέρη του κόσμου αφορά την ανάπτυξη των περιοχών αυτών και το θέμα της σταθερότητας και της πρόσβασης στους πόρους. Σύμφωνα το πρόγραμμα του ΙΕ για το περιβάλλον, 40% των εσωτερικών συγκρούσεων στον κόσμο, εδώ και 60 χρόνια και παραπάνω, εξηγούνται από συγκρούσεις για τα ορυκτά αυτά και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. επικεφαλή της αποστολής του ΙΕ στο Κονγκό λέει ότι θα πρέπει να είναι υπεύθυνε οι επιχειρήσεις και δεν μπορούν να αρκούνται απλώς στην επιχειρηματικότητα και στην εκμετάλλευση των ορυχείων. Πάνω σε αυτή τη δήλωση μπορούμε να βρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντική επιρροή, διότι 28 δισεκατομμύρια των εξαγωγών ορυκτών έχουν προορισμό την Ευρώπη και αν δούμε τις συνιστώσεις των διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούμε, των διαφόρων συσκευών, τις έξυπνες, τα έξυπνα τηλέφωνα, βλέπουμε ότι έχουμε πάνω από 60 δισεκατομμύρια εισαγωγών αυτών των προϊόντων στην ε, Ευρώπη. Έχει μοχλό πίεση η Ευρώπη. Διαβάζοντας το έργο που πραγματοποιήθηκε, μπορούμε να εκφράσουμε μέρη ικανοποίηση για αυτά που έγιναν. Βλέπουμε ότι περιέχονται ενδιαφέροντα στοιχεία στην πρόταση. Εμπνέεται τον οδηγό του ΟΟΣΑ. Ταυτόχρονα έχουμε την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιλέγει ε, μετριοπαθή προσέγγιση. Ε, βήμα-βήμα προσέγγιση. Καμιά φορά αυτό αποτελεί καλή πολιτική. Βλέποντας ότι από το 2010 δεν υπάρχει παρά μόνο πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί την εφαρμογή της αρχής του ΩΣΑ, περίπου 4% των επιχειρήσεων, διερωτώμεθα όσον αφορά την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή εθελοντική εφαρμογή. Και διερωτώμε τι θα ενθαρρύνει τι επιχειρήσεις να συμμορφωθούν οι επιχειρήσεις και να είναι πιο υπεύθυνε στην συμπεριφορά τους. Πάνω από 80 επιχειρήσεις πίστευαν, σύμφωνα με δημοσκόπηση, ότι μόνο μια υποχρεωτική ρύθμιση θα είναι πραγματικά αποτελεσματική. Έχω κάποιες ερωτήσεις λοιπόν. Πρώτο, υποχρεωτικό έναντι εθελοντικού μέτρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτιμά την εθελοντική ε, εφαρμογή διότι υπήρχαν αρνητικοί, αρνητικές συνέπειες στο Κονγκό από την εφαρμογή του νόμου Don't, Don't Frank. Λοιπόν, ήδη το Υπουργείο Ορυχείων της Δημοκρατίας του Κονγκό λέει ότι το επίπεδο της παραγωγής έχει αποκατασταθεί στο κανονικό. Άρα δεν μπλοκαρίστηκε η παραγωγή, ο νόμος Dodd-Frank δημιούργησε μια υπεύθυνη αγορά και έγιναν πολλές πρωτοβουλίες τόπου. Ερώτηση. Η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι επίκαιρη σε σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα, ποιες επιχειρήσεις καλύπτονται. Η εισαγωγή είναι μόνο 0,05 των επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ευρώπη και το Dodd Frank εφαρμόζεται σε όλες τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο στη ΣΥΠΑ. Γιατί δεν έβλεπε υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα των επενδυτών κοινωνίας των πολιτών, ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι φορείς στην διαδικασία της παραγωγής. Τρίτο ερώτημα, τα ορυκτά που αναφέρονται. Ο οδηγός του ΩΣΑ εφαρμόζεται σε όλα τα ορυκτά. Μόνο το προσάρτημα αναφέρεται σε αυτές τις ουσίες. Οι πρώτες ύλες ε, πρέπει κρίσιμες πρώτες ύλες πρέπει να καλύπτονται. Έλεγχοι. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμμετέχει στους ελέγχους. Πέμπτη, προτελευταία ερώτηση. Τα συνοδευτικά μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σειρά συνοδευτικών μέτρων σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκαθαρίσει περαιτέρω τα μέτρα. Τέλος, ορισμός των περιοχών με συγκρούσεις, που αντιμετωπίζουν συγκρούσεις αυτές οι ζώνες συγκρούσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ταυτίζεται με τον ορισμό του ΩΣΑ, άρα να είναι πιο ευρύς ορισμός, πληρέστερος. Γενική βία αναφέρει, ε, παραβιάσεις μάλλον των εθνικών και των διεθνών νόμων ε, είναι ο ορισμός του ΩΣΑ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λούνες έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ. ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα βασιστώ στις σημειώσεις της συναδέλφου που λείπει και για μένα είναι σημαντικό αυτό το θέμα και πιστεύω και εγώ ότι οι προθέσεις του κυρίου Βίνκλερ είναι εξαιρετικές. Όπως είπαν και οι προηγούμενοι, θα ήθελα να αρχίσω αντίθετα από αυτά που είπε η κυρία Αρένα ότι Πρόκειται για ανοιχτό σύστημα και όχι δεσμευτικό και αυτό είναι καλό διότι θεωρούμε ότι μόνο έτσι μπορεί ο ρόλος της Ένωσης να τύχει κάποια εγγύηση, να είναι αξιόπιστος. Αυτό είναι και το μάθημα που πήραμε από το νομοσχέδιο Dodd-Frank. Αλλιώς, θα, αν το σύστημα είναι δεσμευτικό, θα θέσουμε δυσκολίες στους ε, επιχειρηματίες. Λοιπόν, αυτό είναι και το θέμα. Θέλουμε ανοιχτό σύστημα ή μόνο το δεσμευτικό θεωρούμε ότι θα λειτουργήσει. Η πρόταση της Κομισιόν δίνει αρμοδιότητες και στις αρχές των χωρών μελών και τις θέτει στο κέντρο της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτές ας πούμε θα, οι εθνικές αρχές θα αποφασίζουν για τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν τα πιθανά προβλήματα τίθεται βέβαια το πρόβλημα του κατά πόσον θα είναι εγγυημένε αυτές οι απαντήσεις και αντιδράσεις. Και πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, με ποιο τρόπο θα γίνεται ενωσιακά ο έλεγχος. Έχετε κάνει πρώτερη αξιολόγηση του κόστου, τι θα αντιπροσώπευαν όλα αυτά. Έπειτα, θέλω να υποστηρίξω τον κύριο Βίνκλερ το ότι μεγάλο μέρος του νομοθετήματος στοχεύει στην ε, παρεμπόδιση της χρηματοδότησης σειράξεων μέσω της εξαγωγής για μας εισαγωγής τέτοιων ορυκτών. Αλλά νομίζω ότι για να αποφευχθούν σειράξεις χρειάζονται πολύ περισσότεροι πόροι. Το ερώτημα λοιπόν είναι η Κομισιόν εξέτασε τι συμπληρωματικά μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν για την αποφυγή σειράξεων και συμπληρωματικά δεν θα ήταν καλύτερο τέτοια μέτρα να τα να λέει και το κύριο σώμα του νομοθετήματος. Έπειτα η κυρία Αρένα έκανε το διαχωρισμό μεταξύ κυρίαρχων και δευτερευουσών πρώτων υλών. Η χνηλασιμότητα όλων αυτών των υλικών είναι πολύ δύσκολη, αλλά ιδιαίτερα αν θέλουμε να διαχωρίσουμε τις κυριότερες από τις πιο δευτερεύουσες πρώτες ύλε. Δεν ξέρω αν είναι χρήσιμος αυτός ο διαχωρισμός και ίσως θα έπρεπε να λέμε ότι οι δευτερεύουσες πρώτες ύλε δεν θα έπρεπε να αναφέρονται σε αυτόν τον κανονισμό καθόλου. Έπειτα ο ορισμός των περιοχών συγκρούσεων. Είναι και αυτό ο σαφής και εδώ στηρίζω πάλι τον εισηγητή και εγώ νομομαθής και νομίζω ότι ο ορισμός που εφαρμόζεται είναι πολύ ασαφής και στην πράξη θα σήμαινε ότι μπορεί να βρεθούν να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό και χώρες που δεν δικαιολογούν τέτοια θεώρηση ως ζώνες σειράξεων. Ιδίως αν το διευρύνουμε και σε επαπειλούμενες σειράξεις. Δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να κάνει τον κατάλογο αυτών των περιοχών. Τέλος, πρέπει να αποφευχθούν και οι επικαλύψεις. Αν ανεξάρτητη έλεγχοι από ανεξάρτητους οργανισμούς γίνουν για να διαπιστωθεί το κατά πόσον συμβαδίζουν όλα αυτά με τον νόμο Dodd-Frank, τότε ίσως να έπρεπε να δημιουργηθεί ολόκληρο σύστημα πιστοποίησης των πιστοποιήσεων και να χρειάζονται συνεχώς συμπληρωματικοί και όλο και περισσότεροι έλεγχοι. Αν προχωρήσουμε έτσι θα μπορέσουμε να εξετάσουμε κανένα άλλο <clears throat> σημείο της ημέρησης διάταξης. Στις 10 πρέπει να ψηφίσουμε και εκεί πρέπει να σταματήσουμε τη συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν να είστε σύντομοι. Η έκθεση για την Παγκόσμια Τράπεζα θα εξεταστεί μετά από την ψηφοφορία, αλλά τώρα έχουμε μόναχα λίγα λεπτά. Είμαι και Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομη θα προσπαθήσω να είμαι, αλλά μιλώ εξ ονόματο τη Μάρια Δεσάρνε, η οποία είναι αλλά δεν μπορούσε να είναι παρούσα εδώ. Για μα είναι απαραίτητο να δούμε την παγκόσμια δυναμική των ορεικτών από περιοχή ε, σύγκρουση. Είναι σαφέ ότι μπορεί να υπάρξει μια έμεση, άμεση ε, σύνδεση μεταξύ της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων και ένοπλων συγκρούσεων. Η Ευρώπη πρέπει να σπάσει αυτή τη σύνδεση. Μερικά σημεία που μας ενδιαφέρουν τα εξής. Ένα σύστημα ελέγχου το οποίο να είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό. Θα πρέπει να το κάνουμε αυτό, να το εξετάσουμε ε, με αντικειμενικό τρόπο και να δούμε τι συνέπειες έχει ένα σύστημα σαν το Dodd-Frank τα μέτρα τα οποία οδηγούν σε ένα είδο εμπάργκο δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικό. Δεύτερον, οι, τα κάτι μελη πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή πιστοποίηση. Οι εταιρείε θα πρέπει να έχουν μια, μια βοήθεια από τα κράτη-μέλη και κατευθύνσει για το πώ πρέπει να αντιμετωπίζουν το, τον έλεγχο αυτό, το λεγόμενο due diligence. Θα πρέπει οι εταιρείε να ξέρουν πώ τι καλύπτουν. Οι διαδικασίε ελέγχου και υποπτία πρέπει να είναι αποτελεσματικέ. Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι των εισαγωγέων από εθνικές αρχές και ευρωπαϊκές αρχές ή χρειάζεται μονάχα μία αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξασφαλίσει την ισότητα ανταγωνισμού. Και τρίτον, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε εταιρείε οι οποίες ήδη εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου και εποπτείας στην αλυσίδα παραγωγή ε, προμήθειάς τους και θα πρέπει να έχουν συστήματα τα οποία ανταμείβουν τους υπεύθυνους ε, εισαγωγής η αγορά μπορεί να βοηθήσει αυτούς που είναι υπεύθυνοι όπως γίνεται και με την αρχή της εταιρικής ευθύνης. Να το ξέρουν και οι προμηθευτές και οι πελάτες ότι κάποιος είναι υπεύθυνος. Τέλος, τα συστήματα εποπτείας και ελέγχου θα πρέπει να απαρτήσουν τμήμα ενός ευρύτερου πλαισίου που να αντιμετωπίζει τις συγκρούσεις αλλά και να προλαμβάνει τις συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα πρέπει τα σύστηματα αυτά να είναι συμβατά με το αμερικανικό σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1602 της πράξης Dodd Frank και πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να συμμορφωθούν και με τα δύο συστήματα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Πρέπει μακροπρόθεσμα να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι κανόνες θα ενθαρρύνουν και άλλα κρατημέλη να ακολουθήσουν τον ίδιο τρόπο, τον ίδιο δρόμο και εδώ θα πρέπει να βασιστούμε στους εταίρους μας ώστε να υπάρξει μια διεθνής ισότητα ανταγωνισμού και όχι στρεβλώσεις. Το να ξεκινήσουμε με τις δικές μας, αυτό είναι πάρα πολύ λογικό. Να κάνουμε από εκεί την αρχή. Ο Χέλμουτ. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Είναι πολλά αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοί μου, τα οποία μπορώ και εγώ να τα υιοθετήσω. Πιστεύω ότι ευτυχώς η Κομισιόν επιτέλους μας παρουσιάζει μια πρόταση σε σχέση με τον εμπόριο σε ορυκτά που προέρχονται από, περι οχές συγκρούσεων. Πρέπει να πούμε όμω σαφώ και το είπα και διάφοροι συνάδελφοι, ότι δεν είμαστε στην πρωτοπορία. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ήδη την νομοθεσία Dodd-Frank, όπως αναφέρατε προηγουμένω. Και επομένω το τμήμα 1502 ή 1602, επίσης ακόμα και οι Κινέζοι έχουν λάβει κάποια μέτρα για τα ορυκτά από περιοχέ σύγκρουση ή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μια σειρά προτάσει. Ερχόμαστε τελευταίοι και καταϊδρωμένοι κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με αυτή την πρόταση. Έχουμε λοιπόν καλύτερα παραδείγματα για νομοθεσία τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη και από την άποψη αυτή με απογοητεύει η Κομισιόν. Πρέπει να συνεργαστούμε με την Κομισιόν, με τον εισηγητή και όλους τους συναδέλφους για να καταλήξουμε σε ένα σωστό πλαίσιο το πιο σημαντικό για μας είναι να είναι δεσμευτική αυτή η ρύθμιση. Πολλοί συνάδελφοι, πολλές ΜΚΟ λένε ότι το εθελοντικό σύστημα της Κομισιόν δεν πρόκειται να εμποδίσει ορυκτά που έρχονται από περιοχές συγκρούσεων ή παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικαιωμάτων συγγνώμη, να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα είναι επαρκές ένα εθελοντικό σχήμα. 80% από τις 186 επιχειρήσεις που είναι ενεργές στον τομέα αυτό δεν δίνουν καθόλου δημόσιες πληροφορίες για την προέλευση των ορυκτών τους. Και έχω και μία επιστολή από επενδυτικές εταιρείες που έχουν συνολικό τζίρο 800 δισεκατομμύρια δολαρίων που θεωρούν ότι πρέπει να ευθυγραμμιστούν αυτές οι ρυθμίσει στην Ευρώπη με την νομοθεσία Dodd-Frank. Η Κομισιόν επίσης θέλει να περιορίσει το σχήμα αυτό σε πρωτογενείς ε, ε, εταιρείες ε, εισαγωγή και όχι σε μεταγενέστερες εισαγωγέ. Και επίσης δεν καταλαβαίνουμε γιατί πρέπει να περιλαμβάνει μόνο αυτά τα τέσσερα μέταλλα που αναφέρονται εδώ. Υπάρχουν και άλλα ορυκτά τα οποία <clears throat> που προέρχονται ε, από περιοχές συγκρούσεων. Υπάρχει το θέμα της παιδικής εργασίας στη Δυτική Αφρική επίσης και επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ουκρανία που είναι από τις πλουσιότερες πηγές ορυκτών είναι και αυτή μια περιοχή που γίνεται ζώνη συγκρούσεων. Από τη διαδικασία του Kimberley μάθαμε ότι είναι δυνατό να υπάρξει κάποιος έλεγχος του εμπορίου. Μπορούμε να έχουμε τους υπεύθυνου επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένα σωστό ρόλο ώστε να μην χρηματοδοτεί χωρίς να το θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις συγκρούσεις σε άλλα μέρη του κόσμου. Ελπίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την πρόταση ένα αποτελεσματικό μέτωπο για να σταματήσουμε τις συγκρούσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Χέλμουτ και δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειες. Για το υποχρεωτικό τμήμα είναι κρίσιμου σημασία να μην είναι θελοντικό το όλο σύστημα. Το εθελοντικό απεδείχθη αναποτελεσματικό. Και αν θεσπίζουμε ένα νόμο, θέλουμε ένα αποτελεσματικό και μπορεί να λειτουργήσει μόνο υπό υποχρεωτικό καθεστώ. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια παραδείγματα από εταιρείε δεν α, συμμορφώθηκαν με το εθελοντικό σύστημα που ήδη υπάρχει. Με το dodd Frank έχουμε ένα παράδειγμα που πρέπει να μελετήσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Κυρίως αυτοί που ανέφεραν εμπάργκο κλπ. Δείχνουν τα στοιχεία ότι υπάρχει, υπάρχει σημαντικό εμπόριο από τα πιστοποιημένα ορυχεία οι εταιρείε δεν ψάχνουν να βρουν εναλλακτικού προμηθευτέ. Δεν αποτρέπει το εμπόριο καθόλου ο νόμος Dodd-Frank, αλλά βοηθά και συμβάλλει στην ε, αλλαγή την επιτόπια και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε ε, υπόψη και να μάθουμε πώς να βελτιώσουμε την κατάσταση. Δεν πρόκειται για εμπάργκο, αυτό είναι σίγουρο. Και όχι η αποτροπή του εμπορίου. Και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με ένα ανταγωνιστικό σύστημα. Έχουμε το υποχρεωτικό Don Frank. Η χρησιμότητα του εθελοντικού σε άλλους τομείς ε, είναι κάτι που να εξετάσουμε. Δημιουργούμε ένα ανταγωνιστικό σύστημα εδώ που θα δημιουργήσει και προβλήματα. Κανείς δεν ξέρει με τι να συμμορφωθεί τελικά. Και μετά δεν πρέπει ίσως να περιοριστούμε στις πρώτες ύλες, αλλά και στα τελικά προϊόντα για τον καταναλωτή. Είναι σημαντικό οι δεμοί θα αφήσουμε εκτός σημαντικό τμήμα του εμπορίου. Συμφωνώ με τον Χέλμουτ και για το πεδίο των υλικών που καλύπτονται. Αν δούμε άλλα ζητήματα, άνθρακα και ε, χαλκό που προέρχονται από μερικέ συγκρούσεων. Σήμερα θα συζητήσουμε το Μιανμάρ, όπου το θέμα ε, του χρυσού, των ρουμπινιών, και άλλων προϊόντων είναι σημαντικό. Λοιπόν, πρέπει να τα αυτά υπόψη. Και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ομάδα εμπειρογνωμόνων που έχει δημιουργήσει το Συμβούλιο Εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω θα συμμετέχει και ένα μέλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήταν ενδιαφέρον να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Τι είναι αυτή η ομάδα εμπειρογνωμόνων διότι εμείς νομοθετούμε και θα ήταν κρίμα αν κάποια ομάδα εμπειρογνωμών και κλεισμένων των θυρών με συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών, όπως συνήθως γίνεται με ομάδα εμπειρογνωμών... κάνει συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών. Ε, θα ήθελα να ξέρω μέρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ήδη ετοιμάζουν κατευθυντήριες γραμμές, κάποιο εγχειρίδιο περί εφαρμογής του κανονισμού. Πριν έχουμε ψηφίσει, πριν έχουμε καν στα χέρια μας τον κανονισμό. Θα ήθελα διευκρινήσεις ποια είναι η κατάσταση και ελπίζω να μην ετοιμάζετε ένα εγχειρίδιο για κάποιο κανονισμό που δεν υφίσταται ε, καν. Κυρία Μπιγκίνη, ευχαριστώ. Συνάδελφοι, συζητάμε ένα νομοθέτημα πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή την ιδέα της πιστοποίησης για τα ορυκτά που προέρχονται από αίρια συγκρούσεων, κάτι που δεν είναι καινούριο. Εδώ και πολύ χρόνο ε, διαπιστώθηκε ανάγκη γι' αυτή. Δεν μιλώ για το χρή δεν μιλάω για το χρυσό και μόνο, αλλά για το ταντάλιο, το ψευδάργυρο και το βολφράμιο, που είναι πολύ σημαντικά για τα ηλεκτρονικά προϊόντα που εισάγονται σε μεγάλε ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό θέμα, δεν πρέπει να κινηθούμε μόνο ιδεολογικά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα των κατοίκων, των περιοχών και των εργαζομένων που προέρχονται τα Και ταυτόχρονα όμω, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να προσέχουμε να μην δημιουργήσουμε υποβολικό, γραφειοτικό άχθο για τι επιχειρήσει μα που ήδη πλήττονται από την κρίση. Λοιπόν, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, οι Αμερικανοί που τόσο τους επικρίνω όταν ασχολούμαι το TTIP, θέσπισαν μια νομοθεσία πιο προχωρημένη από τη δική μας που εγγυάται η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώνει τι μεγαλύτερε εταιρείε να δικαιολογούν από πού παίρνουν τα μέταλλα που χρησιμοποιούν και είχαν σημαντικά αποτελέσματα κυρίω στο Κογκό. Λοιπόν, σε σύγκριση με την Αμερικανική νομοθεσία, αυτό ο κανονισμό είναι κάπω ε, ε, ρηχό, δεν είναι αποτελεσματικό, είναι ένα πρώτο βήμα αλλά θεσπίζοντα θελοντικό με, ε, μηχανισμό πιστοποίηση, όπως είπαν και οι προελίστες συνάδελφοι ε, δεν νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη λύση και θα εφαρμόζεται μόνο σε αγωγείς, τους άμεσους αγωγείς που πραγματικά είναι ελάχιστοι και όχι σε εκείνους που το χρησιμοποιούν για την παραγωγή προϊόντων. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν εμπνεόμενη εν από την Αμερικανική νομοθεσία να είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας του μέτρου θα πρέπει να γίνονται καλύτεροι ορισμοί όσον αφορά τις περιοχές συγκρούσεων, να αξιολογήσουμε αν πρέπει να επεκταθεί ο κανονισμός για άλλα ορυκτά. Και θα έπρεπε να είναι πιο ευρύ το πεδίο, να μην καλύπτει μόνο τους αγωγή, του άμεσους αγωγείς, αλλά όλη την αλυσίδα παραγωγής και θα πρέπει να προβλέπεται κάποια εξαίρεση για τις μισομεσές επιχειρήσει, διότι το σύστημα για αυτές θα είναι πολύ μεγάλο γραφειοκρατικό άχθος. Ευχαριστώ. So, liebe Δυστυχώς αγαπητοί συνάδελφοι δεν μπορώ να επιτρέψω άλλες παρεμβάσεις διότι ο χρόνος έχει περάσει. Έχουν λοιπόν χρησιμοποιήσει εκπρόσωποι των ομάδων το ημίωρο αυτό για να αναφέρουν τα σημαντικότερα θέματα. Ίσως πρέπει να γίνει συζήτηση περαιτέρω μέσα στα πολιτικά κόμματα για το πώς θέλουμε να προχωρήσουμε. Θα ξαναδώσω για πέντε λεπτά λοιπόν το λόγο στην Κομισιόν για να απαντήσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ερωτήσεις. Δεν περίμενα τόσες. Θα προσπαθήσω να τις ομαδοποιήσω. <clears throat> Καταρχήν, πώς καθορίζουμε τις περιοχές συγκρούσεων. Ας είμαι σαφής στο σημείο αυτό. Η Κομισιόν δεν θέλει να έχει ένα κατάλογο περιοχών συγκρούσεων. Για δύο λόγους αυτό. Πρώτα απ' όλα, το να έχουμε ένα συγκεκριμένο κατάλογο δεν θα είναι αποτελεσματικό. Γιατί οι περιοχές συγκρούσεων αλλάζουν με τον χρόνο. Κάποιες νέες περιοχές εμφανίζονται, κάποιες άλλες περιοχές πάβουν να είναι προβληματικές. Θα πρέπει να γίνεται λοιπόν συνέχεια μία αναθεώρηση κάτι το οποίο είναι δύσκολο και δεν θέλουμε να δώσουμε ένα πολιτικό μήνυμα ότι πρέπει να σκεφτόμαστε μοναχα για περιοχές και χώρες. Γι' αυτό προτιμούμε να αναπτύξουμε και πήρα το μήνυμα από πολλά μέλη που λένε ότι είναι ασαφής ορισμός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς εργαζόμαστε παράλληλα με την νομοθετική διαδικασία για να προετοιμάσουμε πιο συγκεκριμένες κατευθυντήρες γραμμές για να ετοιμάσουμε ένα εγκόλπιο το οποίο θα μπορούσε να βοηθά τις εταιρείες και αυτός είναι ένας μηχανισμός που βασίζεται στις διαδικασίες, επομένως θα πρέπει να εφαρμοστεί από τις εταιρείε αυτές. Προετοιμάσουμε λοιπόν αυτό το εγχειρίδιο, το εγκόλπιο, για να βοηθήσουμε τις εταιρείε να καταλάβουν πού έχουν μία σύγκρουση. Για να έχουμε λοιπόν αυτές τις κατευθυντήρες γραμμές πρέπει να ζητήσουμε και τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων στον τομέα αυτό <clears throat> που θα μας δώσουν τις συμβολές και τα φώτα τους. έρχομαι στο θέμα του εθελοντικού υποχρεωτικού συστήματος που το έφτιαξαν πολλοί ομιλητέ. Η Κομισιόν έχει προτείνει ένα εθελοντικό σύστημα. Αναλύσαμε προηγουμένως τις δύο αυτές εναλλακτικές λύσεις. Θα προσκαλούσα τα μέλη να διαβάσουν την έκθεση αξιολόγησης αντικτύπου και θα δουν ότι έχουμε σταθμίσει όλες τις επιλογές, μεταξύ των οποίων και την επιλογή ενός υποχρεωτικού συστήματος και καταλήξαμε ότι <clears throat> όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα να έχουμε ένα θελοντικό σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό να αποφύγουμε συστήματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις από το να αποχωρήσουν από τις περιοχές σύγκρουσης, όπως έγινε με τον Dodd Frank. Τα προϊόντα για τα οποία μιλάμε εδώ, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, δεν είναι προϊόντα τα οποία παράγονται μόνο στις περιοχές συγκρούσεων. Είναι σημαντική παραγωγή από τις περιοχές συγκρούσεων, μεν, αλλά υπάρχουν Υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες παράγουν τα προϊόντα αυτά και μπορούν οι επιχειρήσεις να βασίζονται σε άλλες περιοχές. Αλλά φυσικά δεν θέλουμε να υποχρεώσουμε τις επιχειρήσεις να αποχωρήσουν πλήρως από τις περιοχές συγκρούσεων. Υπήρξαν και κάποια μέλη του Κοινοβουλίου που είπαν ότι η νομοθεσία Dodd-Frank δεν οδήγησε σε αποχώρηση επιχειρήσεων από την περιοχή των μεγάλων λιμνών. Εδώ έχουμε διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν ότι στην αρχή υπήρξε μια σημαντική μείωση στην παραγωγή ορυκτών από την περιοχή αυτή. Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις και αποκλίνοντα αρνητικά στοιχεία, τα οποία είναι δύσκολο να συμβιβάσει κανείς σε ό,τι αφορά την παραγωγή και τις εξαγωγές από τις χώρες της περιοχής αυτής, αλλά εγώ θα προσκαλούσα τα μέλη μας, τα μέλη της Επιτροπής σας, να δουν την έκθεση <clears throat> των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που εκδίδουν μια αιτήσια έκθεση αξιολόγησης της κατάστασης και για μια σειρά ετών υπογραμμίζουν το γεγονός ότι υπάρχει αντίκτυπος στην παραγωγή, υπάρχει αντίκτυπος στη λαθρεμπορία ορυκτών, γίνεται περισσότερο νόμιμο εμπόριο. Αυτό σημαίνει ότι μειώνονται τα δυνητικά έσοδα για τις χώρες παραγωγής. Και έχουμε επίσης ενδείξεις από μεμονωμένε εταιρείε οι οποίε αποφασίστηκαν, <coughs> συγγνώμη, αποφάσισαν να μην παίρνουν πια ε, ορυκτά από τις περιοχές συγκρούσεων μετά από την έγκριση της νομοθεσίας Dodd Frank. Είναι καλύτερο λοιπόν να είμαστε <coughs> ε, επιφυλακτικοί και να έχουμε μια βαθμία διαδικασία, αυτό το οποίο μετράει και απαντώ σε πολλά μέλη επίσης. Το θέμα είναι πόσοι θα συν, συμμετάσχουν σε αυτό το εθελοντικό σύστημα. Στην αρχική μου παραουσίαση προσπάθησα να εξηγήσω γιατί θεωρούμε ότι θα υπάρξει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που θα δεχτούν αυτό το σύστημα λόγω και της πίεσης των ομοτήμων επειδή είναι και λίγε εταιρείε στο γκεζί αυτό θεωρούμε ότι θα υπάρξει σημαντική συμμετοχή. Και έχουμε συμπεριλάβει στις προτάσεις μας ένα μηχανισμό αναθεώρησης. Μετά από τρία χρόνια θα υπάρξει μια αναθεώρηση και έχουμε αναφέρει ότι αυτή η, αυτή η αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε προτάσεις τροποποίησης του συστήματος από την Κομισιόν και αυτό συμπεριλαμβάνει <clears throat> την συμπερίληψη στοιχείων δεσμευτικού χαρακτήρα. Είναι μια βαθμία λοιπόν διαδικασία. Πιστεύουμε ότι με, τις, ε, τα κίνητρα που δίνονται για τα μεταποιημένα προϊόντα αυτό θα μας επιτρέψει να συμπεριλάβουμε το δυνατόν περισσότερε εταιρείε. Καταλαβαίνω ότι δεν έχετε χρόνο. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Ίσως μπορώ να αντιμετωπίσω τα θέματα αυτά διμερώς. Ναι, θα έχουμε την ακρόαση στην επόμενη συνεδρίασή μας, ίσως διμερώς μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους ε, βουλευτές που θέλουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα. Θέλω πάρα πολύ, κύριε Βίνκλερ, θέλετε να πείτε κάτι. Ξέρω, Πρόεδρε, ότι δεν μπορώ τώρα να συμπληρώσω την ολοκληρώσω, δεν έχουμε χρόνο. Αλλά πρόσεξα όλους ιδιαίτερως τα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ πολύ για τις απόψεις που εκφράστηκαν. Νομίζω ότι μοιάζει θέση μου με αυτή του Πρόεδρου Ομπάμα. Έχασε το Κογκρέσο και είπε ότι έχουμε πολλά κοινά σημεία προς επεξεργασία. Πράγματι υπάρχει κοινό έδαφος για να εργαστούμε. Είμαι πολύ ειλικρινής όταν το λέω. Πρέπει να θυμόμαστε τη δουλειά που έκανε πριν αυτή η Επιτροπή, που είναι Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου του Κοινοβουλίου. Εργαστήκαμε το θέμα για της διαδικασίας Κίμπελη και για άλλα θέματα και πρέπει να θυμόμαστε και τις αποφάσεις μας. Να πω το εξής. Κάτι που είπε ο συνάδελφος. Συντονίστρια της Άλτε. Χρειάζεται αντικειμενική συζήτηση με ανοιχτό πνεύμα. Πράγματι αυτό χρειαζόμαστε. Στη χώρα που ξέρω καλά, κάποιοι λένε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Thanks a lot Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σίγουρος ότι έχουμε ανοιχτό πνεύμα για τη συζήτηση, θα έχουμε ανοιχτό πνεύμα στη συζήτηση και με την ακρόαση στην επόμενη σύνοδο της Επιτροπής. Ευχαριστώ και Βίνκρα, καλή τύχη με τη δουλειά σας. Και έτσι στο τέλος θα έχουμε μια καλή έκθεση που θα την έχουμε στα χέρια μας αρχές του επόμενου έτους. Ξεκινάμε τις ψηφοφορίες, συνάδελφοι. Ελπίζω να έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορίας σας μαζί σας. And we'll start. Zunächst mit der Abstimmung. Πρώτα απ' όλα Δεν ξέρω γιατί έχετε ανεβάσει τα μεγάφωνα αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί καλεσμένοι. Τελείωσε η συζήτηση. Είμαστε τώρα στη φάση της ε, ψηφοφορίας. Παρακαλώ κάντε λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Σημείο 21. Η έγκριση της ανάληψης ε, διαπραγματεύσεων σε σχέση με την συλλογή στατιστικών στοιχείων. Μία και μόνη ψηφοφορία εδώ, άθετη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 32-4 με μεγάλη πλειοψηφία ενεκρίνει. Θα ξεκινήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο λοιπόν. Σημείο 22. Η προφορική ερώτηση για τα προϊόντα διτής χρήσης. Και εδώ έχουμε μοναχαμία ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και εδώ με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Κομισιόν. Σημείο 3, σημείο 23, συγγνώμη. Οι τροποποίησει λόγω της προσχώρησης της Κροατίας και εδώ πάλι έχουμε μία μοναχά ψηφοφορία, άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. με σαρουχική πλειοψηφία εγκρίθηκε αυτό το θέμα. 24. Η ψηφοφορία της γνωμοδότησής μας για τα novel foods, για τα νέα τρόφιμα. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 1, υπέρ. Όχι ηλεκτρονικά, με ανάταση χειρών κανονικά, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Περνάμε στην τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Το μπλοκ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 62 υπέρ κατά άποχες απέριπτε 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε Τροπολογία 67. Έχουμε μια προφορική τροποποίηση. Υπάρχουν αντίρρησεις για την προφορική τροποποίηση. Όχι. Ψηφίζουμε την 67 λοιπόν όπως έχει τροποποιηθεί προφορικά. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Πάλι ηλεκτρικός έλεγχος. 68. Πέρας. Απορρίπτεται όμως η 68. 69. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Για την 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 83. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. 88 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ της 88 κατά αποχές απορρίφθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πάει και αυτό. Απορρίπτεται. 90 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 ψήφι υπέρ κατά αποχές το 93. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 94. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πλοκ 2. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 97. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά δεκτή συγγνώμη, αποχές αποχές για την 100 Α, εντάξει, εγκρίνεται τότε. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτω. 103 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 105 αλλά και 106 που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτή δεκτές. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 29 υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Δεν γίνεται δεκτή. Ξέχασα όμως την τροπολογία συμβιβασμού εξ αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη. Υπέρ, κατά, απόχες, εγκρίνεται. 31. υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. <clears throat> Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Θέλετε έλεγχο. Έλεγχος για την 38. Άρχεται. Πέρας. Στο τσακ πέρασε. Στο τσακ πέρασε. Τριάντα εννιά. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Σαράντα υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται. Άρχεται. Πέρος, πέρας. Με σημαντική πλειοψηφία εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Κίρτον Ντάρλινγκ. Είκοσι Συμφωνία Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Γεωργία, μία μόνο ψηφοφορία ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία και το ψήφισμα σημείο 26 για την Γεωργία και πάλι ξεκινώ με την τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ. Η 11 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστή 2 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε για τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεν εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 21 Συγγνώμη, 20. 20. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Δύο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τελική ψηφοφορία λοιπόν, ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με σαφή πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Ρεν. Τελειώσαμε λοιπόν τις ψηφοφορίες. τελείωσαν οι ψηφοφορίε, πράγματι. Συγχαρητήρια στον κύριο Ρεν. Ναι, τα αποτελέσματα ήταν στον πίνακα. Ξαναγυρίζουμε στο σημείο 20 την παρουσίαση της Παγκόσμιας Τράπεζας. 15 λεπτά είναι ο χρόνος που θα αποδώσουμε στο θέμα αυτό. Λόπες Κλάρος, ο Διευθυντής της Μονάδος για τους ε, Παγκόσμιους Ενδείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας, είναι αυτός ο οποίος θα λάβει το λόγο και θα μας πληροφορήσει για την έκθεση δραστηριοτήτων της Παγκόσμιας Τράπεζας σε ό,τι αφορά το έτος 2015, λέω ο Πρόεδρος και θα μας δώσει κάποιες ενδείξεις για την οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ όσοι θέλουν να φύγουν να το πράξουν και κατά τα άλλα να είναι σιωπηλοί. Συνεχίζουμε το έργο μας, σας παρακαλώ ησυχία στην τάξη. Η εκτιμήση λοιπόν της ε, παγκόσμιας οικονομικής κατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντική για την Επιτροπή μας και γι' αυτό χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Λόπεχ Κλάρος, ο οποίος θα παρουσιάσει την έκθεση αυτή. Παρακαλώ. Καλημέρα Πρόεδρε. Χαίρομαι που εδώ στην Επιτροπή του Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να σας δώσω μια γενική εικόνα των αποτελεσμάτων της εκθέσεως του 2015 για την επιχειρηματικότητα πέρα από την αποδοτικότητα. Θα ήθελα να χωρίσω τα σχόλιά μου σε τρία μέρη, να πω λίγα πράγματα για τις αλλαγές που κάνουμε στην έκθεση Doing Business και πώς θα αλλάξουμε τη μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε. Να σας πω κάποια πράγματα για τα αποτελέσματα της φετινής έκθεσης υπό το φως των αλλαγών και τέλος επειδή αυτή την έκθεση την ετοιμάζουμε επί 12 χρόνια να σας πω ποιες τάσεις διαπιστώνουμε στα στοιχεία. Κάποιες τάσεις είναι αρκετά, μάλλον είναι πολύ ενθαρρυντικές. Η έκθεση αυτή, Doing Business, καλύπτει διάφορες στοιχείες της ε, ποιότητας του περιβάλλοντος επιχειρηματικότητας αντίθετα από την έκθεση περί ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που εξετάζει παραγωγικότητα και άλλους παράγοντες η δική μας έκθεση εστιάζεται επί λίγων τομέων που καλύπτουν ε, κάποιες διαστάσεις των επενδύσεων αν θέλετε να ξέρετε πόσα βήματα, ποιο είναι το χρονικό διάστημα και ποιο το κόστος ε, μιας ε, ΕΠΕ, για τη σύσταση μιας ΕΠΕ, η έκθεση αυτή δίνει τις πληροφορίες. Αν θέλετε να ξέρετε πόσο χρειάζεται ε, για μια σύμβαση, για την καταχώρηση υπηρεσιακών στοιχείων, διασυνοριακό εμπόριο, εισαγωγές, εξαγωγές και ηλεκτρική σύνδεση και καταβολή των φόρων στο κράτος έχουμε κατασκευάσει, έχουμε θεσπίσει κάποιους δείκτες που καλύπτουν όλες αυτές τις διαστάσεις και μάλιστα αποτελεσματικά. Η έκθεση αυτή βασίζεται και στην ερμηνεία εξετάζοντας τον αστικό κώδικα, τον εμπορικό κώδικα, τον φορολογικό κώδικα, ε, των πολιτικών υποθέσεων, περί και, περί, ε, και όλους αυτούς, όλα αυτά τα στοιχεία τα βάζουμε μέσα στους δείκτες. Έχουμε πολλούς δείκτες που εξετάζουν και την επιτόπια κατάσταση. Πόσο χρειάζεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση, πόσο χρόνος χρειάζεται να πληρώσει κανείς τους φόρους του κλπ. Έχουμε πολύ καλό συνδυασμό των νομικών επιταγών και των πραγματικών καταστάσεων. Ε, διαπιστώνουμε ποια είναι η πραγματικότητα. Να σας δείξω μια, κάποιες διαφάνειες που θα σας δείξουν γιατί η έκθεση ήταν τόσο επιτυχής. Εργαλείο για την προώθηση μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις όλο τον κόσμο. Βλέπετε εδώ στο διάγραμμα τι, ποια είναι η κατάσταση για την καταγραφή περιουσιακών στοιχείων στο Βέλγιο. Χρειάζεται 8 διαδικασίες. το ύψος κάθε γραφήματος δείχνει το χρόνο που χρειάζεται η κάθε διαδικασία στο Βέλιο, χρειάζεται 64 μέρες στο ιστόγραμμα και το κόστος είναι 12,7% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που καταχωρείται. Κάτι δαπανηρό, χρονοβόρο και διαδικαστικά δυσχερές. Τα στοιχεία για το Περού τώρα. Τέσσερις διαδικασίες εκεί, 6,5 μέρες, ένα δέκατο του χρόνου που απαιτείται στο Βέλγιο και το κόστος είναι πολύ πιο λογικό. 3,3% της αξίας του περιουσιακού στοιχείου που καταχωρείται. Να πω κάποια πράγματα για τις δύο διαφάνειες. Πρώτον, και είναι χαρακτηριστικό των στοιχείων μας, μπορούμε να σας παρουσιάζουμε όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με συγκεκριμένη συναλλαγή. Σε αυτή την περίπτωση, η καταχώρηση περιουσιακού στοιχείου μπορεί να το κάνουμε αυτό 189 χώρε, να εντοπίσουμε όλε τι διαδικασίε για όλε τι χώρε, για όλα τα έτη, για και έχουμε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας. Όμως, επέλεξα δύο χώρες, Βέλγιο και Περού, σκόπιμα. Α, πριν από 10 χρόνια, αν έκανα την ίδια παρουσίαση εδώ, θα επέλεγα ίσως χώρα του ΟΣΑ, σαν παράδειγμα ταχείας διαδικασίας και εύκολης διαδικασίας. Και θα επέλεγα χώρα του οτισόμενου κόσμου για να δείξω πως τα πράγματα εκεί πηγαίνουν πιο αργά, είναι πιο περίπλοκες διαδικασίες και πιο δαπανηρές. Στο παράδειγμα του Βελγίου και του Περού που επέλεξα, βλέπετε ότι ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Είναι περίπλοκα τα πράγματα, είναι διαδικαστικά δύσκολα και δαπανηρά στο Βέλγιο και σχετικά εύκολα τα πράγματα και γρήγορα στο Περού. Αυτό είναι κάτι που αρχίζει να το διαπιστώνει κανείς βλέποντας τα στοιχεία μας. Θα σας δείξω και άλλες διαφάνειες. Δηλαδή, σε πολλές χώρες του ανατισσόμενου κόσμου οι αρχές υιοθετούν καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές από ό,τι στις χώρες με υψηλότερο εισόδημα. Εδώ, στην έκθεσή μας, τη φετινή, έχουμε 230 μεταρρυθμίσεις που αναφέρονται σε 123 χώρες. και βλέπουμε ότι οι αρχές προσπαθούν να εφαρμόσουν ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων σε όλο τον κόσμο. Ενθαρρυνόμαστε από τα αποτελέσματα στην υποσαχάρια Αφρική. 75 μεταρρυθμίσεις εφαρμόστηκαν στον τελευταίο κύκλο. Άλλη περιοχή πολύ ενδιαφέρουσα. Ευρώπη και Κεντρική Ασία. Εκεί βρίσκονται πολλά μελλοντικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 85% των χωρών εφαρμόζουν μία, δύο ή περισσότερες μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στην έκθεση Doing Business. Κάποιες αλλαγές που έχουμε εφαρμόσει στην έκθεσή μας φέτος μας ικανοποιούν οι αλλαγές. Θεωρούμε ότι θα αυξηθεί η φήμη ε, και η χρησιμότητα της εκθέσεως για όσους διαμορφών πολιτική στον κόσμο. Η έκθεση ταξινομεί τις χώρες, βαθμολογεί σύμφωνα με την νομοθεσία. Δηλαδή έχουμε ταξινόμηση όσον αφορά την ευκολία του επιχειρήν. Το δημοσιεύουμε αυτό κάθε χρόνο. Ένα από τα πράγματα που κάνω τα τελευταια δυο δύο-τρία χρόνια ήταν πειραματισμοί. Με την απόσταση μέχρι τα σύνορα, με ένα νέο παράγοντα που λαμβάνει υπόψη. Μαζέψαμε πάρα πολλά στοιχεία επί δεκαετία για πολλές χώρες και μάθαμε που ακολουθούνται οι καλύτερες ε, πρακτικές για το επιχείρημα. Στην Σιγκαπούρη χρειάζεται κανεί 150 μέρε για να εφαρμόσει μια σύμβαση. Σε πολλέ χώρε χρειάζονται 3, 4, 5, 6, 7, 8 χρόνια, πολύ περισσότερο. Προφανέ αυτό είναι κακό για του επιχειρηματίε. Στη Σιγκαπούρη όμω η καλύτερη πρακτική ακολουθείται στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά την, την εφαρμογή των συμβάσεων, την επιβολή των συμβάσεων το χρόνο είναι στην πρώτη γραμμή η Σιγκαπούρη. Στη Νέα Ζηλανδία χρειάζεται μισή μέρα να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Εκεί είναι τα σύνορα όσον αφορά να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Για όλους τους υποδείκτες και όλους τους δείκτες και τη δειγματοληψία δημιουργήσαμε αυτό το σύνορο με βάση τα στοιχεία. Βλέπετε τις, ε, τα κίτρινα στίγματα στο γράφημα. Για κάθε χώρα σας δείχνουμε πόσο μακριά είναι από τα σύνορα της βέλτιστης ε, πρακτικής όσον αφορά την επιχειρηματική νομοθεσία. Τι θεσπίσαμε φέτος. Χρησιμοποιούμε την απόσταση μέχρι τα σύνορα σαν βάση για τη βαθμολόγηση. Δεν ακολουθούμε πλέον την κλασική ταξινόμηση. Χρησιμοποιούμε την ταξινόμηση που μετρά την απόσταση της χώρας από τα ιδανικά σύνορα. Ε, είναι αρκετά υποφελές αυτό και η παλή μεθοδολογία βαθμολόγησης και η καινούργια ε, συσχετίζονται στενά. Ένα όφελος όμως για, από το να χρησιμοποιούμε το, την τρόπο μέτρησης απόσταση από τα σύνορα είναι στον πίνακα 1-1 το βλέπετε. Πλέον από τη βαθμολόγηση επιπλέον δείχνουμε και τι βαθμό έχει πάρει η χώρα για να, βαθμολο... για να τοποθετηθεί. Και η βαθμολόγηση ομαδοποιείται δεν είναι καταναμημένοι ομοιόμορφα. Στο Περού, Χιλή, Βέλγιο, Ισραήλ, Μεξικό, Κολομβία, όλες αυτές οι χώρες έχουν βαθμούς πολύ παρόμοιους παρόλο που η θέση τους ε, στον πίνακα είναι διαφορετική. Ε, και βλέπετε ε, το βέλος, το γαλάζιο δεξιά. Τι σημαίνει ότι η απόσταση προς τα σύνορα βελτιώθηκε. Έχουν ανωδική πορεία. Και όπως βλέπετε στον πινακα περίπου 80% από τις χώρες έχουν βελτιώσει την απόστασή τους από τα σύνορα και τη σχετική βαθμολόγηση το 2014. Παρόλο που σε πολλές περιπτώσεις ε, να έχασαν, ε, είναι σε χαμηλότερη θέση βαθμολογικά. Αυτό που είναι σημαντικό για τις αρχές είναι η απόσταση από τα σύνορα. Αν έχει βελτιωθεί αυτή, σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον έχει βελτιωθεί και το δείχνουν οι δείχτες μας. Αυτό είναι θαρρυντικό μήνυμα που αποστέλλεται. Μπορούμε να πούμε σε χώρες, 80% των χωρών, ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον φέτος είναι καλύτερο από πέρσι. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Και ο νέος αυτός συντελεστής, ο νέος τρόπος μέτρησης αυτός, αυτός αυτή η νέα παράμετρος είναι πολύ σημαντική γι' αυτό. Κάτι άλλο. Έχουμε επεκτείνει την κάλυψη όσον αφορά τα στοιχεία στις μεγάλες χώρες με πληθυσμό πάνω από 100 εκατομμύρια σε, και καλύπτουμε και δεύτερη πόλη. Είχε ακουστεί κάποια επίκριση κατά τη έκθεση μα κατά το παρελθόν. Μα λέγανε ότι λαμβάνεται υπόψη το επιχειρηματικό περιβάλλον στι μεγαλύτερε ε, πόλει και αυτό ίσω να μην είναι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει σε όλη τη χώρα. Η Ρωσία διαμαρτυρόταν τυπικά. Ε, λέει ότι ασχολείστε με τη Μόσχα, αλλά η Ρωσία έχει πολλές χρονικές ζώνες ε, και υπάρχουν άλλες ε, πόλεις όπου έχουν καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οπότε στην έκθεση Doing Business η Ρωσία παίρνει χειρότερο βαθμό και θέση από ότι αν τα στοιχεία ήταν πιο αντιπροσωπευτικά. Για να καλύψουμε αυτό, αυτή την επίκριση προσπαθήσαμε να επεκταθούμε σε 11 χώρες με πάνω από 100 εκατομμύρια κατοίκους σε δεύτερη πόλη στη ΣΥΠΑ, πέρα της Νέας Υόρκης, βάλαμε και το Λος Άντζελες. Στο Μεξικό Έχουμε το Μοντερέι στη Βραζιλία, έχουμε το Ρίο Τεζανίρο κλπ. στην Ινδία. Πέρα από το Μουμπάι πήγαμε και στο Δελχή, στην Κίνα, πήγαμε από Σανγκάι, Πεκίνο. Βλέπετε στο χάρτη ποια είναι η κάλυψη. Τι ανακαλύψαμε με τα συλλογή των στοιχείων. Για κάποιους δείκτες, οι δείκτες που βασίζονται σε εθνική νομοθεσία δεν βλέπουμε αλλαγή ο νόμος για την προστασία των επενδυτών ή για την ε, πιστο... Ε, απόκτηση πιστώσεων, για την πιστοληψία εξαρτάται από την εθνική νομοθεσία. Οπότε δεν υπάρχει μεταβολή να αλλάξουμε πόλη. Κάποιοι από τους άλλους δείκτες που συνεπάγονται χρονικό στοιχείο, δηλαδή το χρόνο ξεκινήσει επιχείρηση, ο χρόνος να καταγραφεί μια ε, ένα περιουσιακό στοιχείο για την καταβολή των φόρων. Υπάρχει διαφορά μεταξύ δύο πόλεων τη ίδια χώρα. Όπω βλέπετε στη χάρτα στα δεξιά, στο χάρτη στα δεξιά, βλέπουμε τη, τη γραμμή αυτή και δεν υπάρχουν δραματικέ ε, διαφορέ μεταξύ πρώτη και δεύτερη πόλη. Μία εξαίρεση είναι η ΙΠΑ, όπου στο Λος Άντζελες η ποιότητα η επιχειρηματική είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στη Νέα Υόρκη. και η θέση των ΙΠΑ έπεσε κάποιες θέσεις φέτος. Διότι ομαδοποιούμε τα στοιχεία για τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τη θέση της, Νέας της θέσης των ΙΠΑ. Συγγνώμη. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύτερη πόλη ε, δείχνει γενικά, είναι καλή, απεικονίζει αρκετά καλά τη γενική εικόνα της χώρας για το επιχειρηματικό περιβάλλον. Μια-δύο άλλες αλλαγές που κάναμε όσον αφορά την έκθεση και θα κάνουμε φέτος και του χρόνου. Κάνουμε δύο χρόνια μεταρρυθμίσεις. Να σας δώσω κάποια γεύση των αλλαγών. Δύο παραδείγματα να σας δώσω. Το πρώτο. Ο δείκτης για την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Ε, πέρσι ετοιμάσαμε το πρώτο δίκτυο υποδομή, η Παγκόσμια Τράπεζα το ζήτησε αυτό. Ο δείκτης καλύπτει το χρόνο διαδικασίες και το κόστος που αφορούν την σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο. Σημαντικό το, το βήμα για την Παγκόσμια Τράπεζα και για το όλο πρόγραμμα Doing Business και δείχνει ότι ο δείκτης συσχετίζεται με πολλά άλλα θετικά στοιχεία της κοινωνίας. Είναι πολύ καλή εικόνα για την ποιότητα των υποδομών, τουλάχιστον στον ενεργειακό τομέα. Ε, όμως, πολλοί φίλοι μας στην Αφρική, τα, την τελευταία διετία, ήρθαν και μας είπαν, κοιτάξτε, πράγματι είναι πάρα πολύ δαπανηρό να γίνει ηλεκτρική σύνδεση στην Αφρική, αλλά το πραγματικό πρόβλημα εκεί δεν είναι το κόστο τη σύνδεση. το πραγματικό πρόβλημα είναι η αξιοπιστία του εφοδιασμού. Τη στιγμή που συνδεθεί με το δίκτυο πολύ συχνά δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αυτό είναι ο μεγάλο πονοκέφαλος για τον επιχειρηματία που δεν ξέρει πότε θα έχει το ηλεκτρικό ή αν θα έχει ηλεκτρικό όταν το χρειάζεται. Του χρόνου λοιπόν θα προσθέσουμε στο κόστο, διαδικασία και χρόνο για να συνδεθεί κανεί με το ηλεκτρικό δίκτυο και άλλο δίκτυο που θα καλύπτει την αξιοπιστία ε, της ηλεκτρικής παροχής σε 119 χώρες. Πιστεύω ότι ο δείκτης θα αποτελεί βελτίωση, γενική βελτίωση πέρα από τους δείκτες που ήδη έχουμε. Δεύτερο παράδειγμα που σχετίζεται με την καταχώρηση περιουσιακών στοιχείων, περιουσίας. Ο δείκτης ο σχετικός εστιάζεται στην αποτελεσματικότητα διαδικασιών χρόνος, κόστος, διαδικασίες που χρειάζονται για να καταχωρηθεί περιουσιακό στοιχείο από τον πολιτή προς τον αγοραστή ε, εστιάζονται πολύ επί της συναλλαγής. Όμως κάποιοι επικριτές του δίκτυ ήρθαν στην τράπεζα και είπαν «Κοιτάξτε, στη χώρα μας η καταχώρηση περιουσίας χρειάζεται χρόνο, είναι διαδικαστικά περίπλοκο ζήτημα, δαπανηρό, όμως τη στιγμή που θα καταχωρηθεί περιουσία τα δικαιώματα είναι ασφαλή και δεν υπάρχει ε, δικαστική υπόθεση διαμάχη μετά. Σχεδόν ποτέ. Και υπάρχουν κάποιες χώρες όπου είναι πολύ εύκολο να καταχωρηθεί η περιουσία αλλά ίσως η ασφάλεια δικαίου είναι πολύ μικρότερη και υπάρχουν πολλές υποθέσεις στα δικαστήρια. Το θέμα είναι ποιο είναι από καλύτερο, το καλύτερο συστήματα. Αυτές οι επικρίσεις είναι σωστές, αυτό πιστεύω, έχουν κάποιο νόημα. Οπότε αυτό που θα κάνουμε του χρόνου είναι πέρα από το χρόνο, τη διαδικασία και το κόστος της καταχώρησης της περιουσίας θα βάλουμε και ένα δίκτυ που θα καλύπτει διάφορες ποιοτικές διαστάσεις ε, του καθεστώτος για τα περιουσιακά στοιχεία, αξιοπιστία, διαφάνεια, κάλυψη του συστήματος καταχώρησης γεών, διαχείρισης χωροταξικό κλπ. Και μετά θα βάλουμε και ένα ισχυρότερο δίκτυ που θα καλύπτει και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών καθώς και το τι συμβαίνει σε ποιοτικό επίπεδο. Επιτρέψτε μου, κύριε Λόπες, λέει ο Πρόεδρος, χρόνου φίδου. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε σε κάποιες διαφάνειες που δείχνουν τι συμβαίνει σχετικά με τα στοιχεία. Πιο μακροπρόθεσμα. 2005 λοιπόν. Αν διερωτηθείτε σε πόσες χώρες του κόσμου χρειάζεται λιγότερο από 20 μέρες για να ξεκινήσεις μια επιχείρηση, ήταν 20 χώρες, κυρίως του ΟΣΑ. Πληρές χώρες υψηλού εισοδήματος, 2014. Αυτός ο αριθμός αυξήθηκε σε 127 χώρες. Έχουμε κάτι παραπάνω από τριπλασιασμό του αριθμού των χωρών που μπορεί να ξεκινήσει σε μια επιχείρηση σε λιγότερο από 20 ημέρε. Είναι πολύ σημαντικό διότι ξέρουμε από την τεκμηρίωση τη χώρα εκείνε που είναι πιο περίπλοκη κατάσταση για να ξεκινήσει μια επιχείρηση υπάρχουν μεγαλύτερα επίπεδα διαφθορά και παρατυπιών. Τελευταία διαφάνεια, ξέρω ότι μα πιέζει ο χρόνο. Είναι η τελευταία διαφάνεια που σα δείξω όσον αφορά τι μετατροπέ και τι αντιστοιχίε. Αν χωρίσετε το δείγμα και πάνω αριστερά κοιτάξτε στο διάγραμμα της διαφάνειας. Αν χωρίσουμε το δείγμα των χωρών, να δούμε τις χώρες τις χειρότερες που χρειάζονται περισσότερο χρόνο να κάνεις την ετοιμάς την επιχείρηση, τα πράγματα είναι περίπλοκα, δύσκολα και μετά έχουμε τα άλλα, τρια, τα άλλα τμήματα. Μεταξύ 2005 η διαφορά ήταν 87 μέρες του καλύτερου και του χειρότερου. Τώρα μειώθηκε στι 29 μέρε το 2014. Και βλέποντας τι άλλε γραφικέ παραστάσεις υπάρχει σύγκληση ε, των στοιχείων στον κόσμο. Στι χώρε εκείνε που είναι πιο δύσκολη η κατάσταση υιοθετούν καλύτερες πολιτικές και παίρνουν παράδειγμα τι καλύτερε χώρε και για μα την Παγκόσμια Τράπεζα είναι θετικό το μήνυμα, διότι η Παγκόσμια Τράπεζα είναι ένα θεσμό που αφορά συγκλήσει, είναι ένα θεσμό που θέλει να προσπαθήσει να δημιουργήσει στον απτυσσόμενο κόσμο, σε αναπτυσσόμενες χώρες, τις συνθήκες εκείνες που υπάρχουν στις προθυμένες ε, οικονομίες και στην, ε, στις χώρες με υψηλότερο εισόδημα. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτό πράγματι συμβαίνει και είναι πολύ ενθαρρυντικό το μήνυμα που βγαίνει μετά από 10-12 χρόνια της έκθεσης Doing Business. Ευχαριστούμε. Κυρία Δέριν Ντάλιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση από ό,τι καταλαβαίνω εδώ αναμειγνύεται πρακτική με νομικά, με το νομικό πλαίσιο. Στην Αμερική η Κολομβία θεωρείται ως πρώτος εμπορικός εταίρος. Αλλά τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την παραβίασή τους, πώς συμπεριλαμβάνονται αυτά. Σε αντίθεση με το καθαρά νομικό τμήμα. Ηλίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας κύριε Κλάρος και για το πάρα πολύ ενδιαφέρον έργο που έχετε κάνει στα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρώ ότι οι πληροφορίες που δίνετε είναι πάρα πολύ σημαντικές για να καταλαβαίνει κανείς πώς μπορεί να ξεκινήσει μια δραστηριότητα, αλλά δεν έχουμε στοιχεία για την συνέχεια μιας δραστηριότητας από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει στη χώρα μας, παραγωγή χάρη, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ ο δείκτη σε σχέση με την ευκαιρία του να δημιουργήσει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια επιχείρηση. Δεν λέει κανεί όμως τίποτα για τι δυσκολίε που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση για να λειτουργήσει με τη ρύθμιση που είναι όλο και πιο πολύπλοκη και του κανόνε πρέπει να ε, λάβει υπόψη. Δεν ξέρω αν προβλέπετε να εξετάσετε πιο πολύ σε βάθο και αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Μία σύντομη απάντηση, παρακαλώ. Για την Κολομβία, οι ενδείκτε εστιάζονται σε ένα ε, μικρό αριθμό παραγόντων που είναι σημαντικοί για την επιχειρηματικότητα. Δεν, μιλα, δεν εξετάσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση, την ασφάλεια, το επιχειρηματικό κλίμα. Είναι κάπως στενή η οπτική γωνία μας. Αναφέρατε βέβαια το θέμα της ε, ε, ασφάλειας και αυτό δεν περιλαμβάνεται στην έκθεσή μας. Και πρόσφατα η Ισλανδία είχε ένα πολύ καλό δίκτυο για το επιχειρήν, αλλά αυτό συνέβαινε μέσα στην ε, φάση της υποτίμησης του νομίσματος, μια μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση κτλ. Για την ε, ερώτηση της Ισπανίδας συναδελφού, η έρευνα για το επιχειρήν δεν αφορά μονάχα τη δημιουργία μιας επιχείρησης, κοιτάμε και πολλά άλλα στοιχεία μέσα στη ζωή μιας εταιρεία, το να καταγράψει τα στοιχεία του ενεργητικού της, το να πληρώνει φόρους, το να παίρνει άδειες οικοδόμησης, το να αντιμετωπίζει την ε, πτώχευση, το να εφαρμόζει τους όρους ε, συμβολέων, η απόκτηση πιστώσεων κτλ. Είναι πολλοί δείκτε λοιπόν και μόνο ένας δείκτη έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας επιχείρησης. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν όλη την παρουσίαση στους φακέλους μας. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε να σε ξαναδούμε του χρόνου όταν παρουσιάσετε την επόμενη έκθεση. Όλα αυτά είναι πολύ πολύτιμα για το έργο μας στην Επιτροπή ΙΝΤΑ ερχόμαστε στην ε, δημόσια ακρόασή μας για, τις ε, για την επενδυτική συμφωνία με την Μιανμάρ πρώην Βερμανία. Γνωρίζουμε ότι από τότε που ανέλαβε την εξουσία το νέο καθεστώς το 2011 έχουν αλλάξει άρδιν οι συνθήκες στην Μιανμάρ και έχουμε τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις με τη χώρα αυτή και μέσα στο πλαίσιο αυτού του νέου φάσματος δυνατοτήτων έχει παρουσιαστεί μια συμφωνία επενδυτικού χαρακτήρα που θέλει να προωθήσει η Κομισιόν Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ακρόαση. Δεν πρόκειται να κάνω μακροσκελής παρουσιάσεις. Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτά τα οποία μπορούν να μας δώσουν οι καλεσμένοι μας. Προτού τους παρουσιάσω, θα ήθελα να χαιρετήσω την εκπρόσωπο της Υποεπιτρόπης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να τη ζητήσω να μας πει και αυτή κάτι για τα θέματα αυτά, κυρία Λοχμπίλντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Λάγκε. Σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι η Επιτροπή Ίντα έχει προσκαλέσει και την Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποεπιτροπή να είναι παρούσα. Εμείς ως Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πάντα τονίσει την ε, μεγάλη πρόοδο που επετέφθη στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ. Έχουμε στείλει κάποιες αντιπροσωπείες, κάποιες αποστολές στη Μιανμάρ, οι οποίες διαπίστωσαν αυτή την πρόοδο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως Επιτροπή Αρμόδια για τα θέματα αυτά. Μας ενδιαφέρει όχι μόνο η νομοθετική ρύθμιση, αλλά και η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Και βέβαια σε επίπεδο εφαρμογής τα πράγματα δεν πηγαίνουν πολύ καλά. Είναι θετικό το ότι υπάρχει μια Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το θέμα είναι όμως με τι απασχολείται. Αν απασχολείται με μεμονωμένα παράπονα. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι το θέμα των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας γης ή το θέμα της ελευθερίας του τύπου ή η μειονότητα των Ροχίνγκα και η αρπαγή γης στη Μιανμάρ. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εξακολουθούν να λαμβάνουν χώρα στη Μιανμάρ. Ερχόμαστε τώρα σε αυτή τη συμφωνία επενδυτικού χαρακτήρα και εδώ υπάρχει μια ανάγκη να κάνουμε μια αξιολόγηση αντικτύπων στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά έχουμε μονάχα ένα πολύ μικρό κομμάτι μια τέτοια αξιολόγησης. Για μας οι επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσουν τα πρότυπα τα οποία ισχύουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό προβλέπεται να βελτιώσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ. Αυτή είναι η ίδια διατύπωση που ακολουθήθηκε στη συμφωνία με την Κίνα. Αλλά εμείς δεν έχουμε κάποια ένδειξη ότι πράγματι θα γίνει έτσι και γι' αυτό θέλουμε ως Επιτροπή να αντιμετωπίσετε και το θέμα της πραγματικότητας της ε, Μιανμάρ και μέσα στα πλαίσια της ε, εξέτασης αυτής της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιανμάρ θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συνυπολογιστούν. Και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δίνω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο David Martin. Ξέρω ότι δεν έχω χρόνο, θα είμαι σύντομο. Ναι, πράγματι έγιναν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στο Μιανμάρ η εσύ αμφισβητεί κατά πόσο έχει κολλήσει η μεταρρύθμιση και ότι οι αλλαγές ε, που περιμέναμε ότι θα γίνουν δεν γίνονται. Ή τουλάχιστον όχι με τους ρυθμούς ε, που είχαμε πριν από ένα-δύο χρόνια. Επέρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά τα δικαιώματα των μειονοτήτων, κυρίως των μουσουλμάνων, μουσουλμανικής μειονότητας, ε, ε, που δεν έχει αντιμετωπιστεί. Σκοπός της ακρόασης είναι να δούμε πώς μπορούμε να δούμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδυτική συμφωνία με το Μιανμάρ. Πρέπει να εξισορροπήσουμε τις αλλαγές που γίνονται στη χώρα που είναι καλά, ε, στοιχεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ και να το συγκρίνουμε αυτό με τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης. Δεν θέλουμε ευρωπαϊκές εταιρείες να πάνε στο Μιανμάρ και να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, θέλουμε να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκέ εταιρείε που επενδύουν στο Μιανμάρ προστατεύονται παρκώ. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ προστασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με το να εξασφαλίσουμε ότι δεν εκμεταλλευόμαστε στην κατάσταση στο Μιανμάρ. Ευαίσθητη ισορροπία πρέπει να πετύχουμε. Ελπίζουμε ότι η ακρόαση θα συμβάλλει στην εξέβρεση τη ισορροπία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ερχόμαστε στον πρώτο γύρο όπου τίθεται το θέμα της πολιτικής ε, κατάστασης και των επιπτώσεων στο επενδυτικό πλαίσιο της Μιαν. Ε, Κυρία, ο κύριος Όινκ που είναι ο αρμόδιος στο Υπουργείο Εθνικού Σχεδιασμού για τα θέματα αυτά και τα θέματα οικονομικής ανάπτυξης θα μας παρουσιάσει και ο οποίος είναι και ο διαπραγματευτής της Μάς ε, στα θέματα αυτά. Δέκα λεπτά έχετε το χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε πάρα πολύ. Καταρχήν θέλω να σας πω ποιος είμαι. Γενικός Διευθυντής στο τμήμα του Υπουργείου για την Οικονομική Ανάπτυξη και της ε, Επιτροπής Επενδύσεων στην Μιανμάρ. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ και θα ήθελα να σας πω τα τελευταία νέα για τις επενδύσεις στη Μιανμάρ. Θα αρχίσω με μια σύντομη ιστορική παρουσίαση Μιανμάρ βρίσκεται μεταξύ Κίνας και Ινδίας. Έχουμε σύνορα με την Μπαγκλαντές, το Λάος και την Ταϊλάνδη επίσης και η Μιανμάρ είναι λοιπόν μια γέφυρα μεταξύ όλων αυτών των παλαιών εθνών της Νοτιοανατολικής Ασίας. έχει σύνορα και με 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Έχουμε πολλούς φυσικούς πόρους, αλλά δυστυχώς η χώρα μας είναι ακόμη πτωχή. Η αγορά μας είναι μεγάλη, 40 εκατομμύρια. και πάνω από 50-60% του πληθυσμού μας είναι νέοι. Τώρα να σας πω πώς είχε η κατάσταση το 11, ένα χρόνο δηλαδή πριν την ανάληψη της εξουσίας από την καινούργια κυβέρνηση. Το 11 δεν ήταν και τόσο καλά τα πράγματα. Η ανάπτυξη του ΑΕΠ δεν ήταν πολύ υψηλή και το ισοζύγιο πληρωμών επίσης. Ο εξηλεκτρισμός επίσης ήταν πολύ χαμηλός. Η καινούργια κυβέρνηση λοιπόν από τις 30 Μαρτίου του 2011 ανέλαβε πολλές αλλαγές. Οι πρώτες ήταν η μετάβαση από τη στρατιωτική κυβέρνηση στην εκλελεγμένη κυβέρνηση. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στη δημοκρατική μετάβαση. Υπάρχει και μία διαδικασία ειρήνευσης. Η οικονομία μας ήταν ήμι αγοράς και τώρα είναι πλήρους αγοράς. Η κυβέρνηση ανέλαβε πολύ σοβαρές μεταρρυθμίσεις, καταρχήν πολιτικές που βασίστηκαν στην πολιτική ζωή όλων, όλων των πολιτών, στην ελευθεροτυπία και στη συμφιλίωση. Υπήρξαν και προοικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, νέες εμπορικές επενδύσεις και επίση και νομισματικές και δημοσιονομικές αλλαγές. Αυτά τόνισε η κυβέρνησή μας καθώς και μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, όπου βασιστήκαμε κυρίως στην καλή διακυβέρνηση και στην διαφανή και καθαρή διακυβέρνηση. Τέλος, η κυβέρνησή μας θέλησε να αναπτύξει τον ιδιωτικό τομέα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα και τελικά μία μονάδα του Υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε συγκεκριμένα αυτό το τομέα. Αυτές είναι οι κύριες μεταρρυθμίσεις στη Μιανμάρ. για τη δημιουργία του νέου επιχειρησιακού κλίματος καταλάβαμε ότι η ανάπτυξη θα αργήσει, θα είναι μακρόσυρτη η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις όπως την δικαστική μεταρρύθμιση όπου στοχεύουμε μεταξύ άλλων και σε μεγαλύτερη ελκυστικότητα του επενδυτικού κλίματος υπάρχει μεγαλύτερη ελευθέρωση της οικονομίας και υπάρχουν και άλλες πιο διαδικαστικές τεχνικές μεταρρυθμίσεις όπως την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και καλύτερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις. Επίσης θεσμικές μεταρρυθμίσεις η Επιτροπή Επενδύσεων της Μιανμάρ θέλησε να διευκολύνει την οικονομική μετάβαση για όλες τις επιχειρήσεις με συνεργασία όλων των Υπουργείων και η Επενδυτική Επιτροπή αυτή τη στιγμή αποτελείται κατά το ίμιση από υπουργούς και το άλλο μισό από τον ιδιωτικό τομέα οικονομολόγους, προέδρους επιχειρήσεων και μερικοί από το εμπορικό και τεχνικό επιμελητήριο. Αυτά Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να έχουμε ένα ευρύ φάσμα εμπλεκομένων στον τομέα αυτό. Μπορούμε να κάνουμε και μια σύγκρουση μεταξύ του 1998 και του 2011. Η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία Και όπως βλέπετε από το γράφημα αυτό, εάν έχετε υπερμετροπία και το βλέπετε, μπόρεσε να αυξήσει σημαντικά τις επενδύσεις. Ε, το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων είναι στον τομέα της εξόριξης ορυκτών και τότε το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων ήταν στην διαχείριση πρώτων υλών, ενώ τώρα έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος των επενδύσεων στις ε, μεταφορές, στις επικοινωνίες και στην ε, μεταποίηση. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σημαντική αλλαγή στη, των επενδύσεων στην ε, Μιανμάρ, δεν είναι στον εξωτερικό τομέα, αλλά είναι στον τομέα μεταποίησης, στις τηλεπικοινωνίες, σε τομεί υψηλή παραγωγή προστιθέμενη αξία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή μεταξύ τη προηγούμενη κυβέρνηση και τη τωρινή κυβέρνηση. Αν δούμε λοιπόν ε, τι επενδύσει, η Κίνα είναι από τις πιο σημαντικές χώρες οι οποίες κάνουν επενδύσεις στη Μιανμάρ. Ακολουθείται από την Ταϊβάν και την Σιγκαπούρη. Εξακολουθεί η Κίνα να είναι αυτή η οποία κυριαρχεί στις ξένες επενδύσεις στη Μιανμάρ. Και εδώ βλέπετε την αλλαγή, την πρόοδο των επενδύσεων τα χρόνια που έχει αναλάβει την εξουσία η κυβέρνησή μας. Και έχουμε φτάσει σε επίπεδο επενδύσεων 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά έχουμε και 4,3 δισεκατομμύρια που ήρθαν από την Κίνα για σταθμούς ενέργειας και το 2012-2013 οι επενδύσεις φτάσανε τα 1,5 ε, δισεκατομμύρια. Ήταν μια σημαντική λοιπόν αύξηση και τον τρίτο χρόνο 2013-2014 Έχουμε φτάσει στα 4,2 δισεκατομμύρια και εφέτος τους πρώτους έξι μήνες έχουμε περίπου ξεπεράσει μέσα σε έξι μήνες το επίπεδο επενδύσεων από πέρσι. Υπάρχει λοιπόν μια ανωδική πορεία των επενδύσεων στην Μιαμάρ. Αν δούμε τις επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον εξορρυκτικό και μεταποιητικό τομέα είναι σημαντικός εταίρος για τις επενδύσεις στη Μιανμά. Αν δείτε τη σύγκριση μεταξύ του 2011 και του 2014, από το 1% του ΑΕΠ έχει φτάσει στα 7% και οι εξαγωγές έχουν περάσει από 7 δισεκατομμύρια σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια. Επομένως υπάρχει μια σημαντική αύξηση μέσα σε τρία χρόνια και άλλες βελτιώσεις σε άλλους ενδείκτες. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία για τη χώρα μας έχουν βελτιωθεί τα μάλα μέσα στα τρία χρόνια της κυβέρνησής μας. Περιμένουμε λοιπόν περισσότερες επενδύσεις από χώρες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, άλλες ασιατικές χώρες Έχουμε κάνει μια επενδυτική συμφωνία με το Ισραήλ και με το Κουβέιτ και τώρα να σας εξηγήσω γιατί χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας. Γιατί δεν θέλουμε να προωθήσουμε γενικά και αορίστως τις επενδύσεις, θέλουμε επενδύσεις ποιότητος, ε, επενδύσεις οι οποίες βασίζονται στις ε, υπεύθυνε επιχειρήσεις και να έχουμε και μεταλαμπάδευση τεχνολογίας. Θέλουμε να προλάβουμε τις άλλες χώρες και θέλουμε επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας που θα προωθήσουν και την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα μας. Θέλουμε επίσης να εξασφαλίσουμε και την διαφοροποίηση των επενδύσεων, να μην βασιζόμαστε μονάχα σε μία χώρα να επενδύσει στην Μιανμάρ. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ. Περιμένουμε πολύ υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξή της, αλλά θέλουμε τις ε, επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να δημιουργήσουν αμοιβαία ωφέλη μεταξύ των επενδυτών και της χώρας υποδοχής. Η κυβέρνησή μας είναι ήδη δεσμευμένη να προχωρήσει σε επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια συμφωνία επενδυτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και ο Πάρα πολύ συγκεκριμένα και πλήρης ε, πληροφοριών η παρουσίασή σας. Τώρα, έχω τη χαρά να δώσω το λόγο σε περαιτέρω ομιλητές, ο κύριος Τερνέλ από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και την κυρία Χαρτ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε λοιπόν εκπροσώπους του πανεπιστημιακού κόσμου και τον ΜΚΟ που θα αναφερθούν και στο θέμα αυτό. Παρακαλώ κύριε Τουρμό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε για την εισαγωγή και ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο που με κάλεσε να έρθω εδώ από το Σίδνεϊ. Πιστεύω ότι οποιασδήποτε ασυνέπειες, λάθη κλπ. θα θεωρηθούν ότι ανήκουν στη διαφορά του χρόνου, στο jet lag και όχι βάσιμα ε, χαρακτηριστικά του που διαθέτω. Λοιπόν, αυτά που είπε σαν χτες ε, κάπω προετοιμάζουν αυτά που θα πω σήμερα. Είπε και παραθέτω η διεθνής κοινότητα θα βοηθήσει τον καλύτερο τρόπο τη μεταρρυθμιστική διαδικασία αναγνωρίζοντας την κατάσταση στη Βιρμανία για αυτό που είναι. Όχι αυτό που θα θέλαμε να είναι και όχι απλώς ελπίζοντας ότι τα πράγματα θα καταλήξουν αίσια. Όπως είπα, αυτά πρέπει να ακολουθήσουν σήμερα. Ε, αυτό το θέμα ε, είναι και στην καρδιά της μεταρρύθμισης στη Βυρμανία. Ε, στους μεταρρυθμιστές και στο γραφείο του Προέδρου. Αυτή είναι η άποψη. Και αυτή την άποψη θέλω να παρουσιάσω σήμερα και είναι η άποψη που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Δεν αντιπροσωπεύει ε, τον απλό άνθρωπο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Λοιπόν, το πλαίσιο της παρέμβασής μου για την κατάσταση της Βερμανία, για την οικονομία της, είναι το πλαίσιο του 2014. Δεν είναι το πλαίσιο του 2012, όπου εκεί υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία και έκπληξη θα έλεγα για το βαθμό των μεταρρυθμίσεων. Λοιπόν, έτσι ακροθυγώς αναφέρω τις μεταρρυθμίσεις, διότι θα τις αναφέρουμε και θα τις εξετάσουμε, να δούμε πώς τα πήγαν, πώς εφαρμόστηκαν, διότι κατά κάποια έννοια αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Ποιες ήταν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες ξεκίνησαν τον ενθουσιασμό, ποιο ήταν το αίτιο του ενθουσιασμού του 2011 και 2012. Ε, λοιπόν, υπάρχουν κάποια θέματα, πρώτα απ' όλα οι αλλαγέ τη ισοτιμία. Πολλοί εδώ στο Κοινοβούλιο θα θυμούνται ότι η Βερμανία είχε ισοτιμία που κλείδωνε το τζατ, το νόμισμα, 7 τζατ σε ένα δολάριο Αμερικής. Αλλά περίπου τελικά ήταν 1000 τζατ σε, ε, στο δολάριο. Η πραγματική ισοτιμία. Η μεγαλύτερη διαφορά που υπήρξε εκεί, υπήρχε και σοβαρότερη διάσταση πέρα από τη συμβολική διαφορά που έδειχνε το οικονομικό χάος της κατάστασης πρέπει να πούμε, ήταν και ένα όχημα μέσω το οποίο το παλιό καθεστώς τελικά πουλούσε το, το, τον πλούτο των ξένων συναλλάγματος της Βιρμανίας. Δηλαδή τις κρατικές επιχειρήσεις τις έβαλε στα λογιστικά με την παλιά ισοτιμία και όχι με την πραγματική αγοραστική αξία. Και τελικά τσέπωνε τη διαφορά. Η μεταρρύθμιση του 2012, δηλαδή η διακύμανση ελεύθερης διακύμανσης ε, του νομίσματος μας έκανε να προσέχουμε τις μεταρρυθμίσεις στην Βυρμανία. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι κάτι σοβαρό κάνουν, άρα ίσως να κάνουν κάτι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ισοτιμία. Δεύτερον, ο κανόνας, ο νόμος για ξένες επενδύσεις. Ε, τρίτον, παρόμοιοι νόμοι για ειδικέ οικονομικές ζώνες. Τέταρτον, η Κεντρική Τράπεζα, νέος νόμος που θεσπίστηκε για, που έδιναν εξαρτησία στην Κεντρική Τράπεζα και μια σειρά γενικότερων κινήσεων που αφορούσαν το εμπόριο, τον τουρισμό κλπ. Και εκεί ξανά αναφέρθηκα σε κάποιο βαθμό ήδη από τους προλαλήσαντες. Λοιπόν, ακολουθώντας τις μεταρρυθμίσεις το 2011-2012, μετά από αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ε, οι περισσότερες έγιναν την πρώτη διετία και γέμισε με προσδοκίες ο υπόλοιπο κόσμο βλέποντα αυτά. Και τότε θα έλεγα σταμάτησε να προσέχει τι γίνεται στη Βερμανία. Η οικονομία τη Βερμανία σταθεροποιήθηκε, διορθώθηκε, άνοιξε επιχειρηματικά η Βερμανία και στον κόσμο δημιουργήθηκε σύμφωνη γνώμη για την όλη κατάσταση στη Βερμανία. Εδώ λέω ότι αυτή η συνένεση ήταν πρόημη, αυτή η άποψη πρόημη. Και αν δούμε την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που δημιούργησαν την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό ε, θα πρέπει να αρχίσουμε να αμφισβητούμε πολλά από αυτά που θεωρούσαμε σωστά τότε και πιστεύαμε τότε. Θεωρώ ότι το 2014 το παρόν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Βερμανίας είναι επιφανειακό, στενό, ατελές και, και λίγοι λίγο πολύ. Δεν είναι μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει τα πραγματικά αίτια των οικονομικών προβλημάτων της Βερμανίας. Τα περισσότερα προβλήματα πορεύουν που η κυβέρνηση που ασκούσε στενό έλεγχο ε, στα περισσότερα κομμάτια της οικονομίας της χώρας. Η Βερμανία όταν και το 2014 πραγματική οικονομία της αγοράς πεδράζεται επί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων αλλά είναι ελεγχόμενη η οικονομία κρατική. Και ο ιδιωτικό τομέα βασίζεται σε άδειε και χωρίσεις παραχωρήσει που κατά των ε, περιορισμών του κράτου. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο. Οπότε οι μεταρρυθμίσει ε, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά είναι χαλαρώσεις, επεκτάσεις των αδειών και εκχωρήσεων και δεν είναι φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις που ίσως θα θέλαμε να δούμε να εφαρμόζονται. Θα έλεγα επίσης ότι αυτές οι εκτεταμένες άδειε και παραχωρήσεις σε μεγάλο βαθμό, όχι πλήρω, σε μεγάλο βαθμό δόθηκαν ε, σε ψευτοεταιρείες που κυριαρχούν στην, στην οικονομία. Δεν είναι επιχειρηματίες αυτές τις εταιρείες, αλλά ομάδες ε, που είναι κολλητές με την κυβέρνηση. Λοιπόν, βασικός λόγος εξολογήσεως που κάνω, που θεωρώ ότι οι μεταρρυθμίσεις όπως εφαρμόζονται, εφαρμόζονται επιφανειακά και είναι ατελείς. Γιατί το λέω. Οι ίδιες αυτές οι ψευτοεταιρείες που ανήκουν στην κυβέρνηση ε, δένονται με τα συμφέροντα. Δηλαδή, οι αποφάσεις του κράτους επηρεάζονται από τα, τη διαπλοκή. Κάνουν ό,τι μπορούν να αντισταθούν ε, στην φιλελευθερωποίηση να μην χάσουν τα δικαιώματά τους. Ένας φίλος μου λέει για τη Βυρμανία ότι ίσως ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα είναι ένα, δηλαδή παίρνει τη μορφή της οικονομίας του Πούτιν. Και κυριαρχούν οι μπράβοι της κυβέρνησης στην οικονομία. Λοιπόν, το είδαμε με την απόφαση να επιτρεπεί τώρα ε, ξένε τράπεζε να έρθουν στην Βερμανία. Μα εξέπληξε αυτό. Το περιμένουμε μακρόν και πριν από δύο εβδομάδε είπαν ότι εννέα ξένε τράπεζε θα πάρουν άδεια να λειτουργήσουν στη χώρα. Δεν υπήρχαν τράπεζε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω από την Ασία. Μία Αυστραλιανή τράπεζα επίση πετράπη να λειτουργήσει, κυρίω ασιατικέ τράπεζε μπορούν να πάνε. Η κατάσταση νομίζω είναι ένα καλό παράθυρο που μα δείχνει τι γίνεται, διότι οι παραχωρήσει που δόθηκαν στι ξένε τράπεζε ήταν εξαιρετικά περιορισμένε. Οι ξένε τράπεζε μπορούν να δανείσουν μόνο σε αλλοδαπού και ε, ξένε εταιρείε. Μπορούν να δανείσουν σε ξένο νόμισμα. Μπορούν μόνο σε χοντρικέ πωλήσει να αναμειχθούν. Δεν μπορούν να είναι στη λιανική ε, μπορούν να καλύψουν έναν κλάδο τη οικονομία και θα πρέπει να συμμορφώνονται με πάρα πολλέ ε, ρυθμίσει και περιορισμού. Ποιο είναι το πρόβλημα με αυτό. Η Βερμανία είναι μια χώρα που το κεφάλαιο λείπει. Η μία ομάδα που έχει τα κεφάλαια βέβαια είναι αυτά τα συμφέροντα που ανέφερα, της διαπλοκής. Λοιπόν, είναι μικρό κόσμος κάτι, κάποιο πιο σημαντικού είσοδο των ξένων τραπεζών. Είναι μια δυνατότητα για μεγαλύτερο ανταγωνισμό έναντι των συμφερόντων που εχει τα κεφαλαια βεβαια ειναι αυτα τα συμφεροντα που ανεφερα της διαπλοκης λοιπον ειναι μικρο κοσμος καποιο πιο σημαντικου εισοδο των ξενων τραπεζων ειναι μια δυνατοτητα για μεγαλυτερο ανταγωνισμο εναντι των συμφεροντων που προανεφερα Ο οικονομικός τομέας, ο τομέας δεν είναι αυτός ο σκοπός, διευκολύνει το επιχειρήν. Οπότε ε, ε, είναι σοβαρή αυτή η απομόνωση και αποκοπή αυτού του ε, τμήματος της οικονομίας ε, και είναι βέβαια και απώλεια διότι δεν μπορούν να μπουν περισσότερες σύγχρονες τράπεζες στη χώρα. Τώρα πέραν αυτού θα ήθελα να πω ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέχρι τώρα στην πράξη δεν έχουν τηρήσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν το 2011 και το 2012 η αλλαγή της ισοτιμίας Είπα ότι ήταν μια ευκαιρία αυτή που δημιουργήθηκε να διορθωθούν τα λογιστικά της οικονομίας, τα δημοσιονομικά. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Ε, Παραδείγματο χάρη, ε, τα, ε, χάνονται τα έσοδα του φυσικού αερίου της, ε, του Μιανμάρ. Ταρπάζει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομικό Ταμείο, αν εξετάσει κανείς και τα σχετικά λογιστικά θα δει ότι 40% των εισοδημάτων από το αέριο δεν πηγαίνουν στα δημόσια λογιστικά στοιχεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι ακούμε να γίνεται πολλή λόγο για φορολογικέ ε, μεταρρυθμίσει, ε, έλεγχο, διαφάνεια όσον αφορά τα φορολογικά. Αλλά άμα βλέπει κανεί 40% τη πιο σημαντική ε, πηγή εσόδων για την κυβέρνηση, δεν μπαίνει στα λογιστικά. Φαίνεται τελικά ότι αυτό είναι η κορυφή του, του παγόβουνου, ότι όλα τα λεφτά ε, δεν μπαίνουν στα ταμεία. Λοιπόν, για τις επενδύσεις ε, έχουμε εμπόριο, βιομηχανία κλπ. που αναπτύσσεται, αλλά στον εξορυκτικό τομέα έχουμε αλλαγές. Ε, ας πούμε στην ε, κατασκευαστική μεταπητική βιομηχανία δεν βλέπουμε πολλές επενδύσεις, κυρίως στον εξαγωγικό τομέα, που ήταν πάντα πολύ σημαντικό. Ε, λοιπόν, ε, στρατιωτικές δαπάνες είπαν ότι μειώθηκαν στη στην ε, ε, Βυρμανία σαν ποσοστό των γενικών κυβερνητικών δαπανών. Τι συνέβη όμως, ότι κάποια από τα έσοδα μπήκανε με την μία φούσκωσε το μέγεθος του προπολογισμού, δηλαδή το ποσοστό που δίνεται στο στρατό είναι μικρότερο ποσοστό τώρα. Αν δει κανείς απόλυτες δαπάνες, βλέπουμε αύξηση των κυβερνητικών δαπάνων τα τελευταία χρόνια. Την τελευταία διετία οι στατικέ δαπάνε αυξήθηκαν 11%. Για την υγεία οι δαπάνε μειώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια κατά 4%. Συγγνώμη, δεν ομιλητή. Το πρώτο έτος της κυβέρνησης έχει αυξηθεί σημαντικά. Όμως βλέπουμε ότι το περιθώριο μένει παρόμοιο, κυρίως στη φορολογία. Και αυτό έχει συνέπειε η υπονόμευση άλλη μεταρρύθμιση ε, που αφορά την κεντρική τράπεζα. Δηλαδή η κεντρική τράπεζα κανονικά είναι ανεξάρτητη, αλλά βέβαια δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη, διότι το σύστημα το φορολογικό δεν είναι επιτυγμένο, οι δαπάνε είναι παραπάνω από τα έσοδα και μόνο φορέα χρηματοδότηση είναι η κεντρική τράπεζα. Πρέπει να καλύψει το έλλειμμα που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν έχει καμία ανεξαρτησία η τράπεζα κεντρική. Εν τω μεταξύ βέβαια, τελικό τομέα, είναι το θέμα της γεωργίας. Στη γεωργία, ε, η γεωργία είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Η γεωργία ε, αφορά τη ζωή του 70% του πληθυσμού. Ε, και τι συμβαίνει στην Γεωργία. Θα έλεγα ότι δεν έγιναν μεταρρυθμίσεις που έχουν νόημα στην Γεωργία και οι Γεωργοί δεν έχουν βασικές οικονομικές ελευθερίες πώς, τι και πότε να παράγουν. Έχουν ελάχιστο έλεγχο της γης που καλλιεργούν. Λοιπόν, ε, ε, η Ήπεθρος τώρα ε, είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι πριν τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό μπορεί να πει κανείς. Τελικό σχόλιο. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις στη Βυρμανία τελικά έχουν λάβει χώρα. Αυτό είναι αμφισβήτητο Μπορεί να το δει κανείς στους δρόμους της Ραγκούν. Αλλά δεν άγγιξαν την τα θεσμικά όργανα, τα οικονομικά που αρπάζουν τον πλούτο της χώρας και τα δίνουν στους στρατιωτικούς, τους πολιτικούς, στην ελίτ, την πολιτική και τη στρατιωτική. Χρειάζονται θεσμοί για πραγματική μεταρρύθμιση και ολιστική οικονομική ανάπτυξη. Τέτοιοι θεσμοί που εξασφαλίζουν τα δικαιώματα ιδιοκτησία, που δημιουργούν ευκαιρίε και κίνητρα ε, για ανάπτυξη και δημιουργούν κάτι που μοιάζει με κάτος δικαίου, χρειάζονται μια μετάβαση που η Βερμανία ακόμα δεν την έχει ξεκινήσει αυτή τη μετάβαση. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η κυρία Σκότχαρτ. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται και για την τόσο σημαντική αυτή ακρόαση σε μια στιγμή που είναι κρίσιμη για την ιστορία της Βερμανίας. Πέραν αυτών που μόλις ακούσατε, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο ρεαλιστικοί, πιο λογικοί σε σχέση με τις εξελίξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βερμανία, στη Μιανμάρ φέτος. Υπάρχει αυτή η δημοσίευση που είναι διαθέσιμη σε εσά στην είσοδο και παρακολουθεί την πρόοδο που ακολούθησε το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών πέρσι. Αυτό που είδαμε το 2014, ο μεγαλύτερος αριθμός νέων πολιτικών συλλήψεων μετά από τη δημιουργία της, την ανάληψη της εξουσίας από αυτήν την κυβέρνηση. Υπήρξαν πριν από δύο χρόνια πολλά χειροκροτήματα και έπαινη για την πολιτική αλλαγή αλλά έχουμε δει τώρα πάρα πολλούς δημοσιογράφους και εκδότες να πηγαίνουν στη φυλακή. Τον προηγούμενο μήνα ένας δημοσιογράφος ε, έχασε τη ζωή του ενώ ήταν σε κράτηση. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις λοιπόν αυτή τη στιγμή <clears throat> σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό έχει να κάνει και με την επιχειρηματική ε, δραστηριότητα είναι το θέμα της αρπαγής γης και κατάσχεσης γης δημιουργεί μεγαλύτερη ένδια και κάνει ακόμα πιο πιθανή την ανάδυση συγκρούσεων, ιδίως σε περιοχές που μέχρι τώρα δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο συγκρούσεων ή βγαίναν από συγκρούσεις. Πρέπει να αντιμετωπιστεί η ατιμορρησία για να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα ατιμορρησίας. Δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος επίσης σε σχέση με το κράτος δικαίου Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν αυξάνουν τον αρνητικό αντίκτυπο της αρπαγής και κατάσχεσης γη. Η νομοθεσία ακόμα δεν είναι ισοδίκια για όλους τους πολίτες και η διαχείριση και η εφαρμογή των νόμων γίνεται με μεραληπτικό τρόπο. Αυτή η σοβαρή έλλειψη κράτους δικαίου έχει δημιουργήσει μια κατάσταση όπου οι γεωργοί της Μιανμάρ δεν μπορούν να προστατεύσουν την εξουσία τους, την ε, γη τους μάλλον, ή να πάρουν κάποια θεραπεία από το νομικό σύστημα, το δικαστικό σύστημα, και αναγκάζονται να καταφεύγουν στη βία για να προστατεύσουν τις ιδιοκτησίες τους από αυτούς που θέλουν να την αρπάξουν. Μπορεί να θεωρείτε ότι οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αρνητικοί. Έχουμε τώρα ένα θετικό παράδειγμα το οικονομική ζώνη της Τίλαουα. Είναι η βέλτιστη πρακτική αυτή γιατί δεν υπήρξαν φόνοι μέσα σε την περιοχή αυτή με τη συμφωνία της Τίλαουα τα άτομα τα οποία έχουν εκτοπιστεί δια της βίας τους δόθηκαν νέες οικίες που είναι πολύ μικρές. Αυτή η αίθουσα θα μπορούσε να καλύψει έξι τέτοιες ε, κατοικίες είναι τόσο χαμηλό επίπεδου ώστε όταν βρέχει μαζεύουν νερά. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες από τα κουνούπια τα οποία ευνοούνται από τα στάσιμα ύδατα. Δεν μπορούν λοιπόν οι οικογένειες να εξασφαλίσουν την υγεία των παιδιών τους υπήρξαν θέσεις οι οποίες, οι οποίες προσφέρθηκαν σε αυτή την ειδική ζώνη, δηλα, αλλά η καθημερινή, το καθημερινό κόστος ξεπερνάει τα, ε, το ημε, ημερομίσθιο, γιατί είναι 4.000 κιάτ η, ετήσια, η ημερήσια αποζημίωση, αλλά 4.500 το κόστος μεταφοράς. Χάνουν λεφτά δηλαδή οι άνθρωποι όταν δουλεύουν. Έχει υπάρξει αναζωπήρωση των συγκρούσεων. Έχουμε 120.000 ε, εσωτερικά εκτοπισμένους στη Μιανμάρ που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα για να είναι αποδέκτες βοήθειας, ιδίως κοντά στα σύνορα της Κίνας που είναι πολύ κοντά στο οροπέδιο του Θιβέτ και έχουν πολύ σκληρούς χειμώνες. Η βία κατά των γυναικών και η επίθεση εναντίον σχολείων και νοσοκομείων είναι στα σταθερές τακτικές. Και εκεί αυτό αφορά και περιοχές όπου υπήρξαν σχέδια για εκμετάλλευση υδροελεκτικής ε, ενέργειας. Στη δυτική Βυρμανία υπήρχε μια προγενοκτονική κατάσταση πριν από το 2012. Ήταν ακριβώς το πώς παρουσιάστηκε αυτό από την ΕΚΟ και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ. Η κατάσταση αυτή έχει γίνει χειρότερη με το σχέδιο δράσης που εφαρμόστηκε, το οποίο οδηγεί στην μόνιμη, σε ένα μόνιμο διαχωρισμό των μουσουλμάνων από τους άλλους πολίτες Μιανμάρ και οδηγεί στο να κρατώνται σε καταβλισμού, σε στρατόπεδα, ένα εκατομμύριο Ροίγγα. Μόνο το 10% αυτών θα πάρουν ένα είδος πολιτικών δικαιωμάτων που είναι όμως πολιτικά δικαιώματα δεύτερης κατηγορίας με περιορισμένα δικαιώματα στον οικονομικό και πολιτικό τομέα. Οι περισσότερες ενέργειες βίας κατά το Ροχίγκα ακολουθούν ένα σαφές σχήμα. Η βία αυτή έχει σταθεί βολική για να απελευθερώσει γη που χρησιμοποιήθηκε για διάφορα προγράμματα ανάπτυξης. Ενώ αλλού η ειρήνη επανήλθε μετά από πολλά χρόνια συγκρούσεων, βλέπουμε να έχουν ξεκινήσει νέες συγκρούσεις τους τελευταίους μήνες, ιδίως στις περιοχές Μουάν και Κάρεν. Ακόμα και εκεί λοιπόν που είχε υπάρξει κάποια επιτυχία μετά την Ειρηνευτική Συμφωνία, έχουμε νέες συγκρούσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την ε, πρόσβαση στη γη και τους φυσικούς πόρους και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Με αυτό, σε αυτό το χάρτη βλέπετε λοιπόν τις περιοχές αυτές όπου οι δράσεις κατά των μουσουλμάνων και των Ροχίνγκα έχουν φτάσει ένα υψηλό επίπεδο ακροτήτων και πράγματι συμπίπτουν με την αρπαγή γης για διάφορα σχέδια ανάπτυξης. Η Ροχίνγκα είναι από τους πιο καταδιοκόμενους λαούς στον κόσμο και υπόκεινται σε μία σειρά πολιτικών που τώρα γίνονται εθνική νομοθεσία στη Μιανμάρ και θα εφαρμοστούν σε όλους τους μουσουλμάνους του της Μιανμάρ και θα έχουν δυνητικά ε, και επίπτωση σε όλες τις άλλες εθνοτικές μειονότητες που δεν είναι βουδιστές. Αυτό περιλαμβάνει το νόμο για την εθνική προστασία των φυλών που περιλαμβάνει ε, περιορισμούς ποινικοποίηση των μεικτών ε, γάμων, ε, έλεγχος των γεννήσεων για το, ε, για το μουσουλμανικό πληθυσμό. Μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν επίσημα και να εφαρμοστεί στο να μειωθούν τα παιδιά των μουσουλμάνων, περιορισμοί για την πολυγαμία καθώς και για την αλλαγή θρησκείας. Με τον τρόπο αυτό δηλαδή συνεχίζεται αυτό το οποίο θεωρήθηκε στο παρελθόν μια κατάσταση ιονία Απαρτχάιτ. Οι επιχειρήσεις και οι ξένοι επενδυτές είναι τώρα υποπίεση για να κάνουν διακρίσεις εναντίον των μουσουλμάνων και είδα δυνητικούς επενδυτές να μου διαμαρτύρονται ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν αρκεί να μην προσλάβουν μουσουλμάνους. Αρκεί να μην δώσουν συμβόλαια σε επιχειρήσεις που έχουν ιδιοκτήτες μουσουλμάνους. Αν δούμε λοιπόν τις ε, απόψεις ότι η βοήθεια και οι επενδύσεις θα μειώσουν την ε, ένδυα στην Μιανμάρ και θα την οδηγήσουν σε μια πολιτική και οικονομική μετάβαση. Αυτό που βλέπουμε στην πραγματικότητα είναι ότι πολλοί από τους παράγοντες που κάνουν τη χώρα αυτή ένα επικίνδυνο χώρο για επενδύσεις πολιτικά και οικονομικά, οι παράγοντες αυτοί παραμένουν και σε ορισμένε περιπτώσεις έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό το οποίο βλέπουμε επίσης είναι ότι υπάρχει έλλειψη νομικής και θεσμικής μεταρρύθμισης, ώστε οι επενδύσεις αυτές αυξάνουν ουσιαστικά τον κίνδυνο ε, αρπαγής γης, καταστροφής του περιβάλλοντος, σεξουαλικής βίας, απώλειας ζωής, απώλειας περιουσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό λοιπόν και ιδίως δεδομένου ότι η συνολική κατανόηση της κατάστασης στην Μιανμάρ δεν έχει προλάβει τα πρόσφατα γεγονότα και την πραγματικότητα. Πάρα πολλοί λοιπόν βλέπουν ότι το να υπάρξει χώρος για περισσότερες επενδύσεις και εμπόριο ουσιαστικά είναι μια απειλή στα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιβίωση πολλών πολιτών της Μιανμά. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, ανησυχητικό όταν μιλάω σε οργανώσεις βάσης και σε κοινότητες οι οποίες ζουν σε περιοχές σε σύγκρουση τα συγκρουσιακές περιοχές. Ένα από τα θετικά ε, βήματα είναι η πρωτοβουλία για διαφάνεια στον εξοριστικό τομέα που η Βυρμανία έχει ζητήσει να είναι υποψήφια στον τομέα αυτό. Εκεί έχει φανεί ότι υπάρχουν αδύναμοι νόμοι, υπάρχει αδιαφάνεια στις ρυθμίσεις και παρενόχληση της κοινωνίας των πολιτών που θέλει πράγματι να συνταχθεί με τη διαδικασία EITI για τον ε, εξορρυκτικό τομέα και να αυξήσει την ε, συνειδητοποίηση στον τομέα αυτό. Όταν μιλάμε λοιπόν για το αν είναι σκόπιμο να επενδύσει κανείς ή όχι στη Μιανμάρ, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα τις μεταρρυθμίσεις. Εάν δεν γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις για να σταματήσει η ατιμορρησία και να εξασφαλιστεί το κράτος του δικαίου και ιδίως ο σεβασμός και η προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ατόμων, επιχειρήσεων και κοινοτήτων, τότε η παρουσία των επιχειρήσεων από την Ευρώπη θα τις εκθέσει στο κίνδυνο του να εμπλακούν σε σοβαρά διεθνή αδικήματα. Οι εταιρείε αυτές θα είναι πολύ δύσκολο να σεβαστούν τις δικές τους απαιτήσει για σωστό έλεγχο και εξασφάλιση σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές εταιρείε μπορεί να βρουν ότι ο κίνδυνος για τα μελλοντικά τους κέρδη θα είναι πολύ υψηλός, γιατί όταν η Βυρμανία κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, αυτές οι εταιρείε μπορεί να ε, εναχθούν ή θα πρέπει ενδεχομένως να πληρώσουν και το κόστος του ότι μπήκαν βεβαιασμένα στην οικονομία της Μιανμάρ χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στα μέλη για να θέσουν ερωτήματα. Ισκά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις για τις οποίες σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που κάνατε και τον κόπο να έρθετε να μας δείτε. Έχω πολλά ερωτήματα, αλλά βέβαια θα τα θέσω και στην Κομισιόν, γιατί πολύ ενδιαφέρον είναι να ακούσουμε και πώς βλέπει η Κομισιόν τη σύνδεση μεταξύ των συμφωνιών επενδύσεων και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για να δούμε και πώς το θέτουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δίνουμε τα χρήματα με όρους ή όχι την ανθρωπιστική κατάσταση, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ ενδιαφέρον λοιπόν, αλλά αργότερα αυτό θα το δούμε. Θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε το εξής. Η συγκεκριμένη επενδυτική συμφωνία σε σύγκριση με άλλες όπως με τον Καναδά κλπ. Τι νομίζετε ότι θα αλλάξει επιτόπου στην Μιανμάρ. Τι θα αλλάξει για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα μπορούν οι επενδυτές ας πούμε θα έχουν το δικαίωμα να μηνύσουν την κυβέρνηση αν εφαρμοστεί νομοθεσία που να μειώνει τα συμφέροντά τους και τα λοιπά. Ξέρετε τι εννοώ. Επίσης, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχει ήδη κάποια σύνδεση μεταξύ επενδύσεων και χειροτέρεψης της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πώς ερμηνεύεται αυτό πολιτικά, οι επενδύσεις πώς ερμηνεύονται πολιτικά έχουν προτεραιότητα έναντι των δικαιωμάτων ή όχι. Δυστυχώς δεν είναι κανείς άλλος εδώ από τη Μιανμάρ στο δεύτερο γύρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου αν θεωρεί ότι οι προτάσεις της Κομισιόν είναι επαρκής ή αν θεωρεί ότι πρέπει να συμπληρωθούν και από δικές σας. Και αυτό γρήγορα ή όχι. Όλη αυτή η επενδυτική συμφωνία λοιπόν πώς συνδέεται με τις μεταρρυθμίσεις, με την πολιτική κατάσταση, με τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτά. Με ενδιαφέρουν αυτά. Θα ήθελα να ακούσω από τον εκπρόσωπο της Μιανμάρ με ποιο τρόπο οι επενδύσεις θα ε, ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη Μιανμάρ και τι είδους εταιρείε θα ενθαρρύνει. Θα ήθελα επίσης να ξέρω και περισσότερο για την Επιτροπή Επενδύσεων της Μιανμάρ και η οποία μας έχει παρουσιαστεί ως ένας φορέας ο οποίος προστατεύει τον κοινωνικό περίγυρο και το περιβάλλον, αλλά από αυτά που είπε ο κύριος Τάνερς είναι ίσως περισσότερο ένας τρόπος να προστατεύσει τα επενδεδημένα συμφέροντα και να εμποδίσει αυτούς που θέλουν να έρθουν στη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω τα στοιχεία που θα μας παρουσιάσετε εσείς και επίσης αν θεωρείτε ότι υπάρχουν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα οποία εξετάζει η Επιτροπή αυτή, η κυρία Μιούλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προφανώς χαίρομαι πολύ που βλέπω ότι η στρατιωτική κατοχή έληξε στο Μιανμάρ. Χρειάζεται όμως πολύ δουλειά ακόμα. Περιμένουμε κατάπαυση του πυρός σε όλη τη χώρα και να ακολουθήσουν πολιτικές διαπραγματεύσεις. Άκρος εύθραυστη η κατάσταση. Οι επενδύσεις στο Μιανμάρ είναι ευπρόσδεκτες, από ό,τι καταλαβαίνουμε χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είμαι περίεργη για το εξή. Το Μιανμάρ πώς θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντικέ πολιτικές για προστασία των ε, μειονοτήτων θα ισχύσει. Να έχουν ίδιο μερίδιο στην οικονομία. Το ISDS φαίνεται ότι δίνει κάποιες προτιμήσεις στους ξέρους επενδυτές έναντι των τόπιων επενδυτών. Εγώ αναφέρομαι στις μειονότητες, διότι μένουν σε περιοχές οι μειονότητες που έχουν πλούτο πρώτων υλών. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στους ομιλητές για σύντομο, σύντομη παρέμβαση. Α, συγγνώμη, δεν σας είδα που ζητήσατε το λόγο. Ναι, ανησυχώ και ανησυχώ πολύ με αυτά που άκουσα από την παρουσίαση κυρίως όσον αφορά τις μειονότητες. Ε, νομίζω ότι θα, σε οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία με οποιαδήποτε χώρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη σύνταξη αυτής και θα πρέπει να επιμένουμε επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας έκφρασης, της ανεξιθρησκείας. Εάν ε, αρχίσουμε εμπορικές σχέσεις με το Μιανμάρ θα πρέπει αυτά να γίνουν πρώτα πριν συνάψουμε η αδίποτε εμπορική συμφωνία. Νομίζω ότι είναι κατάσταση που προσωμιάζει με αυτή της Νοτιού Αφρικής. Θα πρέπει ε, να μείνει εκτός απομονωμένη η Μιανμάρ μέχρι ότου αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τις ομνότητες. Άκουσα κάτι για έλεγχο γεννήσεων, έλεγχο πληθυσμού. Αυτό είναι φρικτό. Εμείς που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο όπου ε, προστατεύουμε την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πώς μπορούμε καν να διανοούμεθα να μπούμε σε εμπορικέ σχέσεις με τέτοια χώρα. Μέχρι ότου μεταρρυθμιστεί δεν πρέπει να κάνουμε καμία συμφωνία μαζί τους εμπορική. Να δώσω το λόγο τώρα στους τρεις ομιλητές για να απαντήσουν. Ο κύριος Ναϊμ, ο πρώτα, για να απαντήσει. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα, να απαντήσω με τη σειρά τη ο βασικός λόγος για τον οποίο θέλουμε να έχουμε τη συμφωνία επενδυτική με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο εξή. Όπως είπα στην παρουσίασή μου, είναι ότι δεν θέλουμε να βασιστούμε ε, σε, μία, σε λίγες χώρες και στη δική μας χώρα οι επενδύσεις. Θέλουμε να έχουμε πολλές πηγές επενδύσεων, να έρθουν χώρες να επενδύσουν. Καλούμε λοιπόν να επενδύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μιανμάρ είναι πολύ σημαντικό για μας. Θα εξασφαλίσουμε έτσι ότι θα προστατεύονται όλες οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η θέση της κυβέρνησής μας στην έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση για συμφωνία προστασίας των επενδύσεων. Θα είναι ισότιμη η αντιμετώπιση των Ευρωπαίων επενδυτών και άλλων επενδυτών στη χώρα και εθνική, σε εθνικό επίπεδο αντιμετώπιση εξετάζεται. Ε, αυτά έτσι βλέπει το θέμα η κυβέρνηση. Θέλουμε να μην υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον ή κοινωνικές συνέπειες. Όταν δεχτήκαμε την πρόταση, Λάβαμε, ξεκινήσαμε το Υπουργείο για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Ασοκομείας ε, είναι το πρώτο αρμόδιο, δημιουργήθηκε τώρα. Στείλαμε την πρόταση εκεί λοιπόν, στο Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος και Δασοκομείας και... για να δει αν η επένδυση θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Δεύτερον, ζητήσαμε τη συμφωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αν η επένδυση θα δημιουργούσε κάποιες αρνητικές κοινωνικές συνέπειες. Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου και της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν επιτρέπουμε επενδύσεις στο Μιανμάρ. Είναι νέα διαδικασία. Μετά τη θέσπιση του νόμου για ξένες επενδύσεις το 2012, ξεκινήσαμε το 2013 τον προαναφερθέντα μηχανισμό. Θέλουμε οι επενδύσεις να μην έχουν αρνητικές συνέπειες στο περιβάλλον, ούτε στην κοινωνία. Επίσης, και κάτι άλλο. Το αρμόδιο Υπουργείο πάντα εξετάζει την πρόταση, πάει επί τόπου, εκεί που θα γίνει η επένδυση ελέγχει τα πάντα. Έρχεται σε επαφή με την τόπια κοινότητα, ζητάει τα σχόλιά τους. Αν υπάρχει κάτι που δεν δέχεται η τοπική κοινότητα, δεν επιτρέπεται η επένδυση. Ε, κάνουμε τα πάντα, τόσο ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αρνητική συνέπεια για το περιβάλλον και την κοινωνία λόγω της ε, επένδυσης. Ευχαριστώ. Ο αυσταλός ε, ομιλητής μας. Λοιπόν, για τις κακές επενδύσεις που ρωτήσατε και και τι αν μπορεί να παίξει θετικό ρόλο επένδυση ή όχι. Εγώ γιατί ανησυχώ ότι γίνεται σε ένα περιβάλλον όπου το θεσμικό πλαίσιο είναι τέτοιο που μπορεί να χρησιμοποιήσει τις επενδύσεις. Σε κάποιο βαθμό, για κάποιους σαν εμένα που με ενδιαφέρει τι γίνεται στη Μιανμάρ, με ενδιαφέρει περισσότερο πώς θα χρησιμοποιήσει την επένδυση η χώρα. Βλέπουμε στην Ανατολική Ασία ότι αυτό είναι το τυπικό μοντέλο των επενδύσεων ε, οι επενδύσεις ε, βοήθησαν πολύ την Ανατολική Ασία να αναπτυχθεί. Θα μπορούσαν τα πράγματα να εξελιχθούν πολύ θετικά. Θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται, τι θεσμός υπάρχει εντός της Βυρμανίας που μπορεί να δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα για τη χώρα. Υπάρχουν, ε, υπάρχει έλλειψη θεσμών ούτως ώστε να χρησιμοποιηθεί η επένδυση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τώρα το δεύτερο ερώτημα προστατευτικό ε, σύστημα ή προστασία των διαπλεκομένων. Να πω κάτι που είναι καλό. Το MSC είναι το, ένα από τα καλύτερα ιδρύματα στο, στη Μιανμάρ και ο, ο διευθυντής, ο αμμόδιος για τις επενδύσεις ε, προσπαθεί να κάνει τα σωστά πράγματα. Οι διαπλεκόμενοι δεν βρίσκονται στο Υπουργείο αυτό το, το, της χωροταξίας, αλλά από αλλού προέρχονται οι διαπλεκόμενοι. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Είναι διαφορετική πτυχή αυτή των διαπλεκομένων συμφερόντων. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Στόταρτ, ε, ευχαριστώ. Ένα από τα ε, θέματα αφορά την συνοχή των πολιτικών της Ευρώπης. Υπάρχουν δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία, σωστή διακυβέρνηση και αυτά που στεριάζουν με τις ενισχύσεις, τη βοήθεια και τις επενδύσεις. Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση τον Ιούνιο με κάποιον που συνέτασε τη Συμφωνία για την Προστασία των Επενδύσεων. Μου είπε έχουμε μια τυπική ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Του είπα πρέπει να βγείτε εκτό του πλαισίου αυτού εδώ. Χρειαζόμαστε πληρέστατη, λεπτομερέστατη ρήτρα, ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όχι για να προστατεύσουμε απλώ του κατοικού τη χώρα, αλλά για να προστατεύσετε τι εταιρείε σα. Διότι πώ προστατεύετε τι εταιρείε σα από το να βρεθούν σε δυσχερή θέση διότι αρνούνται να κάνουν διακρίσεις κατά των μουσουλμάνων, διότι αρνούνται να παραδιάσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σημαντικό ζήτημα. Σχετικά με το πολιτικό περιβάλλον, αυτό που βλέπουμε είναι προσδοκίες. Προσδοκίες ότι η Ευρώπη και άλλοι βασικοί εμπλεκόμενοι φορείς θα είναι τόσο πρόθυμοι να τρέξουν, να επενδύσουν στη χώρα και να φέρουν τις επιχειρήσεις εντός, που απλώς τυπικά ε, εκφράζουν ανησυχία και φροντίζουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα επιφανειακά. Με μεγάλο κινησμό οι διάφορες αρχές συζητούν το θέμα και στη Βυρμανία και στη νοτιο Ασία. Λένε ναι εντάξει αυτοί οι Ευρωπαίοι όλο κάτι λένε για τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά εντάξει από τη στιγμή που τους αφήσουμε να μιλήσουν να πούνε κάτι θα συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Και γι' αυτό ο πρόεδρος Τιντσέν ε, τον περασμένο μήνα στο Μιλάνο στη, στο Φόρουμ Ευρώπης Ασίας προωθούσε τις επενδύσεις ενώ προσπαθούσε να αποθαρρύνει και να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση από την αναστολή να, να, να αποδυναμωθεί η αναφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα στο ψήφισμα του ΟΗΕ. Θα πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε, έχουμε τον κύριο Μναϊού ο οποίος μπόρεσε να κάνει την αλλαγή από το να είναι στατιωτικός να μπει στην Επιτροπή Επενδύσεων το Μιανμάρ και να κάνει θετικά βήματα προόδου αλλά αυτό δεν αντιστοιχεί με την πραγματικότητα επιτόπια. Έχω πολλούς φοιτητέ που εργάζονται στη βάση, ε, σε επαφή με κοινότητες που πλήττονται σε επίπεδο περιβάλλοντος, από παραβιάσεις του περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και αρπαγής γης και λένε ότι ακόμα και τοπικές κοινότητες, κυρίως από τις μειονότητες, προσπαθούν να επικαλεστούν τοπικούς νόμους που ήδη είναι ε, καταχωρημένοι για την προστασία της περιουσίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμα και τότε διώκονται ακριβώς γι' αυτό. Ακόμα και όταν προσπαθούν να προωθήσουν ε, τον, ε, να χρησιμοποιήσουν τον εθνικό νόμο για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Γι' αυτό έχουμε τον Τιν Τζα, ε, προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που για 13η φορά φυλακίστηκε από τον Ιούνιο, διότι μιλούσε και εκφραζόταν κατά της αρπαγής γης και διερωτάτο γιατί Κάποιες αποφάσεις δικαστηρίων υπέρ τοπικών ε, κοινοτήτων αγνοούνταν και δεν εφαρμοζόταν. Ε, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να δούμε την πραγματικότητα ρεαλιστικά, αντί να παρασυρώμεθα από ρητορικά σχήματα και καλά λόγια. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στον δεύτερο γύρο είναι η επίσημη τώρα, αν θέλετε, άποψη για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε επενδύσεις ε, σε βιώσιμο επίπεδο. Έχουμε τέσσερις σύντομες παρατη... παρουσιάσεις από, την... Ε, από τους οικονομικούς κύκλους, από τα συνδικάτα και την Ευρωπαϊκή Κομισιόν. Ο κ. Μπούμαν, ο οποίος έχει μια μικρή επιχείρηση κλωστοϊφαντουργικών στην περιοχή. Μέλη του Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Νομίζω ότι η Επιτροπή. Ευχαριστώ την Επιτροπή με κάλεσε να μιλήσω εδώ στην Ακρόαση. Καλούμε σαν μέλο τη Ένωση Ξένου Εμπορίου, μια επιχειρηματική οργάνωση που εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Λιανεμπόριο, για να παρουσιάσω τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς σχεδιάζουν επενδύσεις στο Μιανμάρ και πώς θα μπορούσαμε να δώσουμε πρακτικά παραδείγματα από τη χρειαστή εταιρεία μου. Η Paul Group που είναι στην Ολλανδία παράγει παλτά, ζακέτες στο, στην Κίνα, στο Μιανμάρ και στο Βιετνάμ. Έχουμε εργοστάσεις στο Βιετνάμ. Το, ε, ε είναι ίσο, έχει ε, ε, έγκριση ίσο. Απασχολούμε 550 άτομα και σαν επιχείρηση αναγνωρίζουμε το δυναμικό που έχει η Μιανμάρ όταν μάλιστα είδαμε την αλλαγή προς πιο δημοκρατικό σύστημα και αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για επενδύσεις στο Μιανμάρ. Το 2013 ξεκινήσαμε δοκιμαστική φάση αγοράζοντας από ντόπιου παραγωγούς Μιανμάρ και ευρωπαίους πελάτες και δώσαμε στους παραγωγούς υποστήριξη στη διαχείριση, στήριξη τεχνική και σε άλλες Η χώρα προσφέρει πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες και αναπτύσσεται τάχιστα. Βλέπουμε όμως μεγάλους εμπορικούς, ακόμα υπάρχουν εμπορικοί φραγμοί ε, και έχουμε τρεις ομάδες εμπόδιων. Πολιτικά εμπόδια, κοινωνικά εμπόδια, επιχειρηματικά εμπόδια, νομικά εμπόδια. Τώρα σχετικά όσον αφορά τα πολιτικά και κοινωνικά εμπόδια, ε, λαμβάνοντα υπόψη παρουσιάσεις πρώτε παρουσιάσει, θα είμαι σύντομο και θα περιοριστώ αναφέροντα ότι για τι επιχειρήσει για να μπουν σε πειρασμό, να επενδύσουν και να μπορέσουν να ευημερήσουν, χρειάζεται σταθερό, αξιόπιστο και προβλέψιμο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Δυστυχώς το παρόν υπάρχει πολιτική αβεβαιότητα εν ώψη των επικειμένων εκλογών και υπάρχει εθνοτική αναταραχή και αποθαρρύνονται οι σοβαρές, Σοβαρέ ανησυχίε για βιωσιμότητα υπάρχουν, διότι δεν υπάρχει ε, ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα αναγκαία πρότυπα. Και πολύ συχνά δημιουργείται, υπάρχει κίνδυνος για κακή φήμη, γιατί πολύ, υπάρχει πολύ μικρή προστασία για του εργαζομένου, για τα εμπόδια τη επιχειρήση. Ε, είναι κοινά τα εμπόδια για μια αναπτυσσόμενη χώρα. Οι αρχέ του Μιανμάρ εργάζονται σκληρά προ βελτίωση, αλλά το καθήκον του είναι τεράστιο γιατί παραμένουν πάρα πολλά εμπόδια και προκλήσει. Οπότε οι μεταρρυθμίσεις του Μιανμάρ, όπως λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, χρειάζονται κατεπηγόντω σε διάφορου τομεί κυρίω όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, γη, ηλεκτροδότηση και ε, εργάτες με δεξιότητες. Είναι απαραίτητα για να υπάρχει ένα σωστό και δίκαιο διαφανές περιβάλλον περιβαλλοντικό όπου όλε οι επιχειρήσει που να δημιουργήσουν θέσει απασχόληση αναπτυχθούν. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τράπεζα. Αν δώσω παραδείγματα εμποδίων, το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η πρόσβαση στη γη. Μία μη ρεαλιστική και εκδοσκόπο αγορά δημιουργήθηκε από μικρό αριθμό επιχειρηματιών που ευνοήθηκαν από γνώση όσον αφορά τι υποδομέ, τα σχέδια και τι γλώσσε. Καμιά φορά είναι τριπλάσιε ε, οι τιμέ των εδαφών από τι γειτονικέ χώρε. Οι υποδομέ είναι φτωχέ. Ε, λοιπόν, Μπορεί να χρειαστεί δύο ώρες ε, να πας από πόλη σε πόλη, να πας στην Ήπεθρο. Ε, λοιπόν και τελικά μπορεί να κάνεις μέρες γιατί κολλάς στην κίνηση. Το διαδίκτυο είναι περιορισμένο, ε, δεν είναι αξιόπιστο και πολύ συχνά κόβεται το ηλεκτρικό. Δεν υπάρχει αποτελεσματική και διαφανής χρηματοδότηση και οικονομικό περιβάλλον για τη στήριξη των επιχειρήσεων. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε πιστώσεις και κεφάλαιο. Και δεν υπάρχουν μισθωτικά ε, προϊόντα. Λοιπόν, ε, υπάρχει, γίνονται πεζικές συναλλαγές μέσω ε, διαδικτύου, αλλά χρειάζονται εξάμεινο μέχρι να γίνουν. Και διασυνοριακά εμβάσματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δοθούν. Ε, δεν υπάρχουν εκπαιδευμένοι εργάτες, ε, δεν υπάρχει επαρκής σχολική εκπαίδευση και κατάρτιση. Η παραγωγικότητα είναι πολύ χαμηλή στα ντόπια εργοστάσια με αποτέλεσμα μη ρεαλιστικό, ε, μη ρεαλιστικό κόστο εργατικό σε σχέση με γειτονικέ χώρε. Δεν υπάρχει διαθέσιμη τοπική αλυσίδα εφοδιασμού. Όλα τα προϊόντα πρέπει να εισαχθούν. Άρα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία στα σύνορα, εμπόδια και χρειάζεται και χρόνο, χρονοβόρη διαδικασία. Και δεν υπάρχουν ισότιμε συνθήκε. Οι ασιατικοί κατασκευαστέ έχουν επενδύσει και επενδύουν, βλέπετε, ε, με την υποστήριξη των εθνικών ε, κυβερνήσεων. Υπάρχουν και νομικά εμπόδια. Ναι, οι νόμοι εφαρμόζονται, αλλά πολύ συχνά Υπάρχουν πολλοί νόμοι παράλληλα που δημιουργούν χάος και προβλήματα ερμηνεία και λείπει το δικαστικό πλαίσιο. Υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ νομοθεσιών. Οι ντόπιοι νόμοι εξακολουθούν να είναι ξεπερασμένοι, δεν αντιστοιχούν στις διεθνείς προδιαγραφές. Ε, λοιπόν, όπου υπάρχουν νόμοι που αντίκουν ε, πληρούν τι προδιαγραφέ διεθνεί, υπάρχει διαφορά μεταξύ του στόχου του νόμου και τη πρακτική εφαρμογή αυτού. Να δώσω παράδειγμα για δημιουργία μια εταιρεία στη Σιγκαπούρη, με το κάνει σε λίγε μέρε και χρειάζεται ένα εξάμεινο στην ε, Μιανμάρ. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά, ε, πολλέ διευθύνσει που αναμειγνύονται και όλα είναι πολύ απογοητευτικά. Μετά την καταχώρηση επιχειρήση, εξακολουθεί να μην μπορεί να λειτουργήσει, διότι άδεια για να γίνει κάτι τέτοιο μπορεί να απορριφθεί, να καθυστερήσει για να προστατευτούν τα τοπικά συμφέροντα. Η νομική προστασία είναι πολύ χαμηλή και το νομικό σύστημα είναι ανώριμο. Δύσκολο τελικά να προσφύγει σε δικαστήριο και να είναι δίκαιη απόφαση. Διότι τελικά ευνοούνται οι ντόπιοι φορεί. Ε, ετοιμάζεται νέο νόμο για τη θέση των διαφορών, αλλά υπάρχει δυνατότητα ακόμα παρέμβαση των τοπίων. Και θα είναι δύσκολο να λυθούν τα προβλήματα χωρίς να υπάρχει σωστό ε, πλαίσιο νομικό που να επιτρέπει την αναγνώριση και ε, ε να λαμβάνουν υπόψη οι διευθύνσει που Το εργατικό δίκαιο δημιουργεί σύγχυση, 19 διαφορετικοί νόμοι είναι σχετικοί, είναι ασαφείς ε, και υπάρχουν αντιφάσεις σε πολλά σημεία. Οπότε οι αρχές απαντούν με ερωτήσεις και δεν υπάρχει συνέπεια. Ακόμα και το ILO, οι κυβέρνηση Μιανμάρ, ε, οι οργανώσεις της Μιανμάρ, αν τους ρωτήσεις δεν σου δίνουν σαφείς απαντήσεις. Οι αρχέ παίρνουν σοβαρά το θέμα τη παιδική εργασία. Έχει αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Όμω η επαλήθευση, η εξακρίβωση, η σωστή τη ηλικία ακόμα δεν θέσιμη. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα. Το Μιαν εν ευθέτω χρόνο είναι καλή ευκαιρία για ευρωπαϊκό εμπόριο ε, στην περιοχή τη Ασία. Αυτό πιστεύουμε. Η συνεργασία θα είναι υποφελή και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μιανμάρ. Πολιτικά, κοινωνικά και εμπορικά, αλλά θα πρέπει να το προσκύνουν σωστό, οι συνθήκε να είναι σωστέ τα ωφέλη που αναμένονται από μια συμφωνία η προστασία των επενδύσεων θα είναι ότι με τη συμφωνία θα καταλήξει σε επιχειρήσεις να αγνοήσουν τις επιφυλάξεις διότι αισθανθούν προστατευμένες και υποστηριγμένες για να ξεκινήσουν επενδύσεις. Και αυτή η στήριξη θα θέλουμε και δικαστήριο που θα συμμορφώνει τις αρχές του ΟΗΕ και να είναι σωστές οι διαδικασίες, να εφαρμόζονται αυτές, να αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται οι διεθνεί νόμοι Χρειάζονται ισότιμες συνθήκες για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Θέλουμε να υπάρχει και σωστή αγορά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Να δημιουργηθεί αγορά για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις υπηρεσίες. Βασική ανησυχία ποια είναι, ότι κάποια ωφέλη δεν θα ληφθούν υπόψη επαρκώ και θα ληφθεί, χρειαστεί πολλή χρόνο να καταλήξουμε μια συμφωνία και οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα μείνουν πολύ πιο πίσω σε σύγκριση με του Ασιάτε ανταγωνιστέ του. Η Μιανμάρ θα ωφεληθεί από μια τέτοια συμφωνία, διότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα ακολουθούν μακροπρόθεσμη ολιστική προσέγγιση. Και η συμφωνία θα είναι κίνητρο για του ευρωπαίου επενδυτέ να έρθουν στο Μιανμάρ. Και επειδή οι ευρωπαϊκέ επενδύσει θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη της χώρας και του λαού της. Λοιπόν, καταλήγω. Συστήνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί προς διμερή επενδυτική συμφωνία που θα βελτιώσει την, νομική, την ασφάλεια δικαίου στους επενδυτές και θα, ε, επίσης θα ενθαρρύνει προγράμματα του ιδιωτικού τομέα. Αυτή η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά το ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτέ είναι σε δυσχερή θέση σε σχέση με του ανταγωνιστέ του τη Ασία. Οι ασιατικοί, οι ασιάτε παραγωγοί κυριαρχούν στην αγορά τη Μιανμάρ και θα χάσει περαιτέρω έδαφο η Ευρώπη αν δεν υπογράψει σύμφωνα μια συμφωνία σύντομα. Η διμερή συμφωνία θα οδηγήσει σε πιο ισότιμε συνθήκε. Και συστήνω λοιπόν στι αρχέ του Μιανμάρ να εφαρμόσουν σωστά του νόμου, να δημιουργήσουν πολύ ταχύτερα συστήματα, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να στηρίξει του επενδυτέ, να υπάρχει μια θηρίδα για τι άδειε για το κεφάλαιο και για τη γη σε λογικές τιμές. Εξίσου σημαντικό είναι να, ξεκινήσει, ε, να ξεκινήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για να τροφοδοτηθούν ε, οι ανάγκες με ε, εργάτες με δεξιότητες. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορέσει να δημιουργηθεί η βιομηχανία και τέλος συστήνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει στις αρχές της Μιανμάρ στήριξη για να δημιουργηθεί σωστή νομική βάση για τις επενδύσεις. Να ετοιμαστεί το κατάλληλο πλαίσιο με κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των νομοθεσιών. Σωστή εφαρμογή θα ζωντανέψει τη συμφωνία, θα βοηθήσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θα τις κάνει να έρθουν στο Μιανμάρ και να υποστηρίξουν κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τα μάλα, λέει ο για τις εμπειρίες που μα έχετε παρουσιάσει και τι προτάσεις σας. Δίνω το λόγο τώρα στον Όλαντ Φερστάφεν, τον πρόεδρο της ε, Επιτροπής για το Εμπόριο από το Business Europe. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μάρτιν συνάδελφοι, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να προσέλθω. Μιλώ ως εκπρόσωπος του Business Europe και της Διεθνούς του Επιτροπής για τις Επιχειρήσεις. Συνεννοούμαστε με όλες τις χώρες του κόσμου βλέπω. Θα σας πω μερικά πράγματα γιατί είμαι και στέλεχος κάποιας επιχείρησης της Heineken που είναι μια παγκόσμια ζηθοβιομηχανία και αυτή τη στιγμή εγκαθίσταται στη Μιανμάρ. Τι συζητήσαμε στο Business Group, το ξέρετε φυσικά, το ξέρετε. Ε, συνδυάζει πολλές άλλες οργανώσεις. Θα σας πω γιατί η Business Europe θεωρεί ότι από το 2011 έχει αρχίσει να υπάρχει μια θετική ορμή στη Μιανμαρ, όπως και με αυτήν την επενδυτική συμφωνία. Συμφωνεί και το Business Europe με αυτό. And I hope that President Obama... Ελπίζω ο πρόεδρος Ομπάμα και οι άλλοι ηγέτες που θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα να δώσουν και αυτοί το σωστό μήνυμα να ενθαρρυνθούν οι επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στη Βυρμανία όπως εμείς. Βέβαια υπάρχουν πολλά θέματα. Πολλά. Μπορούμε να τα ονομάσουμε φραγμούς, εγώ όμως τα λέω προκλήσεις. Οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να το ξέρουν, αλλά θέλω να σας πω ότι όταν μια επιχείρηση σαν τη δική μας εκτιμά αν πρέπει να επενδύσει ή όχι σε μια χώρα, τρεις επιλογές έχει. Πρώτον, οι φραγμή και οι προκλήσεις να είναι τόσο μεγάλοι ώστε να μην θέλει να επενδύσει και να περιμένει απλώς. Δεύτερη επιλογή, περίπτωση μάλλον, να είναι τόσο μεγάλες οι προκλήσεις που δεν θα λυθούν ποτέ και να μην γίνει η επένδυση. My colleague has referred to here for small... Και η τρίτη επιλογή και για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για μεγάλες, αν πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος είναι διαχειρίσιμος και ότι καλύτερα είναι να πάμε και να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες, τότε να επενδύσουμε. Η εταιρεία μου πήγε στη Μιανμάρ, ήταν στη Μιανμάρ πριν από 10 χρόνια ήδη. Φύγαμε όμως. Λόγω των πιέσεων που που αντιμετωπίζαμε. Πιστεύουμε όμως ότι τώρα η Μιανμάρ είναι στο σωστό δρόμο. Δεν θέλω να, αντι... να αντιμιλήσω με όλους όσους μίλησαν για προβλήματα, γιατί υπάρχουν προβλήματα και μεγάλα. Χρειάζονται ας πούμε υποδομές που δεν υπάρχουν. Το τοπικό εργατικό δυναμικό και η εκπαίδευσή του σε χώρες σαν τη Μιανμάρ θέλουμε να εργαστούμε τοπικά και άρα να βοηθήσουμε και στην εκπαίδευση των ανθρώπων εκεί ώστε να μπορούμε να τους προσλάβουμε. Αυτό είναι το επιχειρησιακό πρότυπο όλων των εταιριών που ξέρω που βρίσκονται στην Μιανμάρ. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. E Νομίζω ότι οι επενδυτικέ ε, συμφωνίες με την Ένωση πρέπει να χρηματοδοτούν τέτοια μετεκπαιδευτικά προγράμματα και οι εταιρείε να δημιουργούν εμορφωτικά κέντρα. Υπάρχουν πολιτικά προβλήματα με τις, στα προγράμματα της κυβέρνησης. Ναι, φυσικά. Και στην Ινδία το έχω δει αυτό. Η Ινδία είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατίες του κόσμου αλλά και η μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Πολλές χώρες λοιπόν έχουν τεράστια γραφειοκρατία. Και εδώ στις Βρυξέλλες υπάρχει γραφειοκρατία. Ορίστε κύριε Λάγκε να μας τα πείτε. Το νομικό πλαίσιο δεν είναι σαφές και αυτό σωστό είναι. Το είδαμε και αυτό ως πρόβλημα χτίζοντας, οικοδομώντας, δημιουργώντας τη ζηθοποιία μας. Υπάρχουν λοιπόν αληθινά προβλήματα. Οι πολιτικοί κίνδυνοι υπάρχουν, υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά και εμείς είμαστε παρόντες εκεί. Και σας βεβαιώνω ότι μια εταιρεία όταν αποφασίζει αν θα επενδύσει δεν χρησιμοποιεί ένα κριτήριο και μόνο, αλλιώς δεν θα πήγαινε κανείς ποτέ στη Ρωσία. Και εμείς είμαστε παρόντες και στη Ρωσία. Έχουμε προβλήματα και στη Ρωσία. Βεβαίω, Όταν πήγα πέρυσι δύο φορές στη Μιανμάρ, συνάντησα για την τιμή να συναντήσω τον πρόεδρο και την Άουν Κι. Καταπληκτική κυρία. Μου μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και μου είπε όμως ότι δεν της αρέσει και η μπύρα. Και είπε παρακαλώ διασφαλίστε ότι ο λαός μου, έτσι λέει ο λαός μου, θα πίνει υπεύθυνα το προϊόν σας. Και βεβαίως έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Δεν υπάρχουν ακόμα οι συνθήκες της ζεφοποσίας στη Μιανμάρ. Να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση του γιατί είναι σημαντικό οι ευρωπαϊκές εταιρείες να εξετάσουν, να αξιολογήσουν τον κίνδυνο τον επιχειρηματικό και τις ευκαιρίες. Εμείς θα μείνουμε εκεί για καιρό. Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες ιστοποιίες στην ε, Ασία εκτός από την Κίνα. Πιστεύουμε ότι από επιχειρηματική άποψη η Μιανμάρ μπορεί να είναι στην ίδια χωρία χωρών όπως με το Βιετνάμ και άλλες χώρες. Δεν βλέπουμε τι θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Όχι, κοιτάμε τι θα γίνει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Αυτή η συμφωνία επενδύσεων είναι κομβικού χαρακτήρα. Θα ήθελα να παροτρύνω τον κύριο Λάγκεν στο σημείο αυτό γιατί προβλεπόταν να γίνει μια Συμβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης Μιανμάρ. Αυτό θα ήταν ένας πολύ καλός χώρος για να συζητήσουμε όλες τις ε, προκλήσεις που έχουμε με τις τοπικές εταιρείες. Γιατί να πάνε οι ευρωπαϊκές εταιρείες, μα κοιτάξτε τι κάνει η Κίνα. Μας παίρνει την πύρα από το στόμα μας. Επενδύει δισεκατομμύρια. Πολύ μεγαλύτερα ποσά από ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες και η Ευρώπη. Αν το δείτε από ανταγωνιστική έποψη, είναι κέριο, είναι κομβικό οι ευρωπαϊκές εταιρείες να ατενίσουν την Μιανμάρ. Εγώ έχω μιλήσει σε πάρα πολλούς για τη δική μου εταιρεία. Δεν μπορώ να τους πείσω, πρέπει να κάνουν τη δική τους αξιολόγηση. Αλλά μην ξεχάσετε ποιος βρίσκεται στη Μιανμάρ. Η General Electric, η Coca-Cola, η Unilever, μου λένε ότι η Unilever βρίσκεται στο προσκήνιο όλων των θεμάτων που μας απασχολήσουν. Το να δουλεύουμε τις τοπικές κοινότητες, ανθρώπινα δικαιώματα, η εταιρική υπευθυνότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι να είναι μια τόσο μεγάλη εταιρική. Η δική μας αντιμετώπιση είναι ναι, επενδύουμε περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Θα εργαστούμε με τους αγρότες, με τους μεροκαματιάριδες. Έτσι μπορεί κανείς να δείξει στην κυβέρνηση, όπως και σε άλλες χώρες, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επιχειρηματικό πλαίσιο. Θα εργαστούμε με τους ε, αγρότες για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το ρύζι για την πύρα μας. Δημιουργούμε σχέδια για εκπαίδευση σε κοινοτικό επίπεδο. Θέλουμε να βοηθήσουμε την ασφάλεια των δρόμων και την υπεύθυνη κατανάλωση μπύρας. Άλλες εταιρείε κάνουν άλλα πράγματα. Αλλά εμείς θέλουμε να το κάνουμε υπεύθυνα γιατί έτσι μπορεί να δείξει κανείς πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επηρεάσουν το κοινωνικό, επιχειρηματικό και νομικό πλαίσιο. Έχουμε προβλήματα, αλλά είναι το, στο πρώτο τρίμηνο του 2015 θα είναι έτοιμο το εργοστάσιό μα Όσοι είσαστε στη Μιαμάρ, ελάτε να τα πιούμε. Θα κλείσω εδώ γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν ερωτήματα και είμαι έτοιμο να τα απαντήσω. Σας ευχαριστούμε για την εντυπωσιακή σας ομιλία. Τώρα, από την πλευρά της, των συνδικαλιστών, ο κύριος Τζέφρι Φόκτ, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος από την Διεθνή Ένωση Εργατικών Ενώσεων. Σας ευχαριστώ που με φέρατε ενώπιον της Επιτροπής σας. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη αυτή η συζήτηση έχουν αρθεί πολλοί περιορισμοί για το εμπόριο και τις επενδύσεις και υπάρχει πολύ ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Μιανμάρ από πολυεθνικές επιχειρήσεις από την Ευρώπη, την Αμερική και την Ασία φυσικά. Η χώρα γιατί τώρα είναι τόσο ελκυστική. Θεωρείτε... Λοιπόν, οι εργάτες πληρώνονται πολύ χαμηλά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες στην ε, Ασία Σύντομα όμω Μιανμάρ θα μπορεί να συναγωνιστεί με άλλη χώρα που έχει φθηνά εργατικά χέρια όπως είναι το Μπαγκλαντέ. Ήδη κάθε μέρα βλέπουμε ότι οι κατασκευαστέ σε άλλα μέρη της Ασίας ε, που εκεί έχουν αυξηθεί τα απειλούν ή θέλουν να φύγουν και να πάνε στο Μιανμάρ. Ε, και στις βιομηχανικές ζώνες που αναπτύσσονται στη χώρα. Μεγάλες εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, ήδη ανακοίνωσαν ότι ενδιαφέρονται να επενδύσουν ή να εμπορευθούν. οι Carlsberg, οι Χάινεκεν το έχουν κάνει ήδη. British American ε, Tobacco, η Ericsson, η Philips, η Statoil, η Mercedes-Benz κλπ. Λοιπόν, η ITUC θέλει να γίνουν επενδύσεις στο Μιανμάρ οι επενδύσει τη Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα δημιουργηθεί νέες θέσεις απασχόλησης, κάτι που χρειάζεται και ανάπτυξη δεξιοτήτων και θα είναι μια αναβάθμιση για τους εργαζόμενους στο Μιανμάρ. Όμως ελλείψη δέσμευση για μεταρρύθμιση, συνοχή σε κοινωνική μεταρρύθμιση και οικονομική μεταρρύθμιση θα πρέπει να γίνει προσπάθεια να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ποιότητα τη απασχόληση που θα δημιουργηθεί δεν σίγουρα θα είναι αξιοπρεπή αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και αν δεν υπάρχουν κατάλληλοι κανόνε. Σίγουρα έγινε πρόοδο για τα εργατικά δικαιώματα. Το είδαμε αυτό, γίνεται προσπάθεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εξακολουθούν υπάρχουν προβλήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και υπάρχει προβληματισμό αν γίνονται πραγματικέ μεταρρυθμίσει. Το 2011-2012 ε, λοιπόν, ε, θεσπίστηκαν νομοσχέδια τη θέση διαφορών και το κρατικό δέκιο και για πρώτη φορά έχουν καταχωρηθεί τα συνδικάτα. Πολύ πρόσδεκτο. Υπάρχουν αυτοί οι νόμοι που είναι λυπεί. περιορίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικάτων και πρέπει να γίνουν αλλαγές. Ε, ε, λοιπόν, υπάρχουν εμπόδια για τους εργαζόμενους στο τοπικό εθνικό επίπεδο. Παραβιάζονται τα εργατικά δικαιώματα σύμφωνα με, το, με τη διεθνή νομοθεσία. Λοιπόν, η οικονομική... υπάρχει φορέας για τα οικονομικά θέματα υπό τον έλεγχο των συντηρητικών στο Μιανμάρ. Χάλιβας, ζάχαρη κλπ. σε αυτούς τους τομείς δεν επιτράπει στους ελεγκτές εργασίας να επισκεφθούν στις μονάδες να δουν αν ο ελάχιστος αριθμός των εργατών ε, υπάρχει για να δημιουργηθεί συνδικάτο, οπότε οι εργάτες θέλουν να μπουν σε συνδικάτο, αλλά δεν τους επιτρέπεται το Υπουργείο Άμυνας διατείνεται ότι είναι εκτός ε, του, της νομοθεσίας, είναι παράνομο κάτι τέτοιο. Η κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την Ομοσπονδία των Συνδικάτων, το Μιανμάρ και άλλες ενώσεις συνδικάτων και έτσι οι εργάτε δεν έχουν φωνή σε εθνικό επίπεδο τη δυνατότητα να μπουν σε τριμερή κοινωνικό διάλογο που είναι σωστό. Και λένε ότι ε, υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, το εργατικό δίκαιο δεν προστατεύει ε, τη συμμετοχή των εργαζομένων στα συνδικάτα ε, και οι ηγέτες των συνδικάτων αφαιρούνται με διάφορες κατηγορίες για κακή συμπεριφορά και κατηγορούνται, μάλιστα απειλούνται με ποινικά δικήματα αν δεν παραιτηθούν. Λοιπόν, η δυνατότητα επιλύσεως των διαφορών ε, και αποφάσεις των δικαστηρίων αγνοούνται ατιμωρητοί. Αν κάποιος δεν σέβεται συμφωνίες ή ε, αποφάσεις διατητικές, ε, ο νόμος αποδυναμώθηκε. 500 δολάρια είναι η μέγιστη ποινή. Δεν είναι κάτι αποτρεπτικό οποιαδήποτε αποτρεπτικο η επιχειρηση καταναγκαστική εργασία, εργασία παιδιών, ε, κατασχέσεις, ε, υποχρεωτικός εκτοπισμός, ε, καταναγκαστικός εκτοπισμός γίνονται στην Βυρμανία. Αυτές οι πρακτικές θα επηρεάσουν και το διεθνή εφοδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να είναι υπεύθυνε κοινωνικά όταν επενδύουν ή εμπορεύονται με το Μιανμάρ. 15 Ιουνίου 2012 οι επίτροποι Άστον και Δεγκούχτ ζήτησαν υπεύθυνε επενδύσεις στο διμερές εμπόριο είναι κάτι σημαντικό για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της χώρας. Και το ίδιο είχε πει το Συμβούλιο τον Απρίλιο 2013 ότι μελλοντικέ δραστηριότητε επενδυτικέ και εμπορικέ από ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θα πρέπει να προωθούν την πρακτική τη ακαιρεότητα και κοινωνική ευθύνη αναφέρεται αυτό στις κατευθυντικές γραμμές του ΟΣΑ για πολυεθνικές εταιρείες. Τις αρχές του ΟΗΕ και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όμως δεν είδαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα να, δώσει, ε, να εφαρμόσει αυτά που έλεγε. Η ΗΠΑ ηγούνται όσον αφορά τις υπεύθυνες επενδύσεις. Έχουν νέες απαιτήσει για τις υπεύθυνες επενδύσεις στη Βερμανία. Οι εταιρείε αμερικανικές ετησίως δημοσία πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρήσεις τους στη Βερμανία, τις συναλλαγές τους, πληρωμές προς κυβερνητικούς φορείς, δικαιώματα ανθρώπινα, καταπολέμηση διαφθοράς, ε, περιβαλλοντικές ε, πολιτικές διαδικασίες. Και το Υπουργείο Οικονομικών τον ΗΠΑ επικαιροποιεί και δημοσιεύει ε, λίστα ατόμων των οποίων τα συμφέροντα και οι διοκτησίες ε, μπλοκάρονται και εμποδίζονται και έχει επικαιροποιηθεί, επικαιροποιείται τακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις τους να συμμορφώνονται με ίδιες προδιαγραφές όπως είπα όταν πηγαίνουν στις, ε, στο Μιανμάρ. Η ITUC πιστεύει ότι όσοι κινούνται επιχειρηματικά εκεί πρέπει να συμμορφώνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να είναι διαφανείς όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Χρειάζεται λογοδοσία, χρειάζεται διαφάνεια. Και πρέπει να υπάρξουν εργαλεία να εφαρμόζονται αρχές του ΟΗΕ και κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ η χώρα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται απόλυτα με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να διορθωθούν τα προβλήματα για να γίνουν επενδύσει. Πρέπει να υπάρχει μηχανισμός διευθετήσεων των διαφορών και υποβολής αναφορών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έτσι δεν θα συμβάλλουν σε αύξηση των προβλημάτων νέες επενδύσεις. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν και κινούνται στη Βερμανία πρέπει να δεχτούν την ανάγκη να κινούνται ανοιχτά και να συνεργάζονται και με τα συνδικάτα μεταξύ άλλων. Παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση του Μιανμάρ να βελτιώσει το εργατικό δίκαιο και να εφαρμόζει το εργατικό δίκαιο. Τέτοιε απαιτήσει είναι προπόθεση για επενδύσει. Θέλουμε προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε βελτίωση των προβλημάτων, λύση του. Και να, έτσι θα μειωθούν και οι κίνδυνοι του επενδυτέ. Θα πρέπει και οι επενδυτέ να στηρίξουν αυτέ τι απαιτήσει με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλουν σωστή ανάπτυξη της Μιανμάρ. Άρα θα δημιουργηθούν αλυσιδωτά και περαιτέρω ευκαιρίες για εταιρείε. Θα... θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν ε, κατάλληλοι κανόνες. Η ITUC συμφωνεί με τις ανησυχίες του ETUC όσον αφορά το περιεχόμενο των επενδυτικών συμφωνιών που προτείνονται. Έχουμε κάνει επικρίσεις και αναφέρθηκαν στο ψήφισμα του ETUC του 2013 για επενδυτική πολιτική. Συζητείται και το θέμα του TTIP και του CTIP και θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προχωρήσει σε διμερείς επενδύσεις που, και, συμφωνίε και συμφωνίες που αντιγράφουν παλιές συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβει υπόψη η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ανησυχίες των ψηφισμάτων που έχουν ψηφιστεί και τα 500 δημόσια σχόλια που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα του TTIP να ληφθούν υπόψη. Θα πρέπει να υπάρξουν σωστοί μηχανισμοί για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη λογοδοσία και αυτά είναι κρισίμου σημασία για δίποτε συμφωνία με το Μιανμάρ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πλήρη εικόνα, πληρέστατη εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο να μας εξηγήσει τι συμπέρασμα μπορεί να συναγάγει από όλα αυτά κ. Κώστα, υποδιευθυντής της αρμόδιας μονάδας για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας όλοι. Η σημερινή μας συζήτηση έθιξε πολλά θέματα και θα ήθελα σήμερα να σας περιγράψω πού ακριβώς βρισκόμαστε και λίγο το ιστορικό του γιατί αποφασίσαμε να κάνουμε μια τέτοια συμφωνία επενδυτική προστασία των επενδύσεων στη Βερμανία. Όπως ακούσατε και το πρωί από τις μαρτυρίες επιχειρήσεων, η Βερμανία έχει δυναμικό, μεγάλο δυναμικό για ανάπτυξη, δυνατότητες ανάπτυξιακές, αλλά και κοινωνικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ε, υπευθύνων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Και εμεί θέλουμε να είμαστε παρόντες στην αγορά της Βερμανίας. Υπάρχουν και ανταγωνιστές μας στην Ασία. Έχουν συναυθεί και άλλες συμφωνίες εκτός από τη Βερμανία με άλλες χώρες του ΑΣΕΑΝ ας πούμε. Η όλη συζήτηση και οι παρουσιάσεις για την ασταθή πολιτική κατάσταση στη Βερμανία σημαίνει ότι η σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας εγγύησης των επενδύσεων είναι ακόμη πιο απαραίτητη διότι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και μετριοπαθείς ως προς το τι μπορεί να καταφέρει μια τέτοια επενδυτική συμφωνία. Τέτοιες συμφωνίες διασφαλίζουν ότι οι επενδυτές που έχουν ήδη επενδύσει σε μια τρίτη χώρα θα προστατεύονται κατά τριών στοιχείων. Άνησης μεταχείρισης, άδικης μεταχείρισης, δηλαδή χωρίς πρόσβαση στη δικαιοσύνη κλπ. Και ε, αποζημίωση σε περίπτωση εθνικοποίησης ή άλλης κατάσχεσης. Δεν γίνεται όμως λόγος για τη δυνατότητα της ε, κυβέρνησης της Βερμανίας να διευθετεί τα πάντα ως προς το πώς θα γίνονται οι επενδύσεις. Θέτουν ορισμένους όρους που και εμείς το μόνο που ζητάμε είναι τους τρεις όρους που αναφέραμε πιο πριν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να διαπραγματευτεί τέτοια συμφωνία με βάση ανάλογες συμφωνίες του παρελθόντος. Και γιατί αυτό, διότι πάντοτε λέγαμε ότι η προσέγγιση μας για τις επενδυτικές συμφωνίες στοχεύει πάντοτε την προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα και αφήνει ελεύθερη την ε, χώρα της επένδυσης να διευθετήσει τα επενδυτικά της. Έχουμε συμφωνίες και με τη Σιγκαπούρη και με τον Καναδά και πάντοτε αποσαφηνίζουμε ποια είναι η φύση και οι όροι, τι εννοούμε δίκαια μεταχείριση, τι εννοούμε κατάσχεση που πρέπει να τύχει αποζημίωσης κλπ. Οι διαδικασίες του ISDS θα γίνουν γνωστές και, και στο ευρύ κοινό. Άρα θα πρόκειται για μία μοντέρνα επενδυτική συμφωνία στη Βερμανία που θα διασφαλίζει και θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που όπως ξέρετε και με την ΕΖΕΣΤΟ συζητάμε. Βέβαια εδώ πρόκειται για μία μεμονωμένη επενδυτική συμφωνία και όχι με αγενική συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Το επεξεργαζόμαστε λοιπόν και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό το θέμα και το κείμενο που θα υποβάλουμε προς τη Βερμανία θα μιλάει για όλα αυτά τα θέματα. Γενικά θα μπορούσα να σας πω ότι οι επενδύσεις θα βοηθήσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη Βερμανία και θα βοηθήσει και τις ευρωπαϊκές εταιρείες να λειτουργήσουν σε αυτό το ασταθές περιβάλλον Πιστεύουμε δε ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα προσφέρουν πολλά στην χώρα αυτή. Ταυτόχρονα η συμφωνία θα είναι όπως είπα πριν μοντέρνα και δεν θα παρεμβαίνει υπερβολικά στις δικαιοδοσίες και τα δικαιώματα της κυβέρνησης της Βερμανίας. Έτσι θα υπάρχει μία αμοιβαία, αμοιβαίως συμφέρουσα συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος τι ακριβώς θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιγράψατε πολλά, αλλά τι γίνεται με τις λεπτομέρειες. Οι λεπτομέρειες μου φάνηκαν κάπως θολές. Ίσως αυτό ήταν κάτι αναμενόμενο. Λοιπόν, η συζήτηση πάει στους συναδέλφους David και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα ακολουθήσουν. Ο Λόδος του Ντάρτμουθ έχει το λόγο. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ, Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα. Θεώρησα ότι ακούσουμε το σύνθημα τη Χάινεκεν. Ότι αναζωογονεί μέρη τα οποία άλλε μπύρε δεν μπορούν καν να αγγίξουν. Πίστεψα ότι θα το πείτε αυτό και για το Μιανμάρ αλλά ενδιαφέροντα τα επενδυτικά σας σχέδια εκεί. Το ερώτημά μου, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν η επενδυτική συμφωνία θέλουμε να έχει κάποια χρησιμότητα πέρα από την προστασία των ευρωπαϊκών επενδύσεων, θα πρέπει να περιέχει και διάλογο και έλεγχο που θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται και από τη δική μας πλευρά θα παρακολουθούμε τη συμπεριφορά ευρωπαϊκών εταιριών που λειτουργούν στη Μιανμάρ και θα είμαστε διάλογο μαζί τους κατά για το πώς λειτουργούν στη Μιανμάρ και όπως είπε και εκπρόσωπος των συνδικάτων αυτό ζήτησε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ψήφισμα που συνέγραψα. Θέλουμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν, ελέγχονται οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές και άλλες προδιαγραφές σε συνάρτηση με τη συμπεριφορά των επιχειρήσεών μας. Απ' την άλλη πλευρά και τώρα με την ίδια τη Μιανμάρ θέλουμε να έχουμε μαζί της ε, διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια συμφωνίας. Γίνονται τακτικά συζητήσεις για τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μιανμάρ αν αυτά τα στοιχεία δεν συμπεριλαμβάνονται απλώς να βελτιώνουμε την προστασία επενδύσεων για τις εταιρείες της ευρωπαϊκές δεν αρκεί. Το επιχείρημα ότι η Κίνα εκεί είναι ήδη και πρέπει να πάει και η Ευρώπη αφού είναι εκεί η Κίνα, κατά την άποψή μου δεν έχει καμία ισχύ εκτός, αν πούμε, ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα βελτιώσει την κατάσταση στην Μιανμάρ, υποθέτοντας βέβαια ότι εμείς συμπεριφερόμαστε καλύτερα και ότι εκεί θα βελτιώσουμε την κατάσταση μέσω του τρόπου με τον οποίο δραστηριοποιούμεθα. Τώρα, τι Δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι επειδή είμαστε Ευρωπαίοι συμπεριφερόμεθα καλύτερα από τους Κινέζους. Αλλά πρέπει να συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λόγω της επικότητας των δύο από τους φιλοξενούμενους θα μιλήσω Ολλανδικά. Πρόεδρε, ε, αναφέρθηκαν όλες οι δυνατότητες που προσφέρονται από τη Μιανμάρ. Εγώ θα ήθελα όμως ε, να ακούσω και κάποιο ντόπιο επιχειρηματία να ξέρω τι γίνεται. Ε, υπάρχουν κάποιοι που υπέγραψαν μια αναφορά, ένα αίτημα κατά αυτής της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αναφέρθηκε η κοινωνία των πολιτών στη Μιανμάρ Πρέπει να τους ακούμε. Εγώ ανησυχώ για την ευάλωτη αυτή δημοκρατία στο Μιανμάρ που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Αν αφήσουμε τώρα στα χέρια των μεγάλων επιχειρήσεων τη χώρα, διαρωτώ με αν αυτό θα είναι προ όφελο των κατοίκων. Έχω δύο ερωτήσει να απευθύνω προς τον κύριο Πούλμαν και τον κύριο Βεστάπεν. Θέλετε να προστατευτείτε κατά των ντόπιων πολιτικών. Αυτό είπε ο κύριο Πούλμαν. Διότι πολλά πράγματα πηγαίνουν στραβά αν, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές οι πτυχές σε συμφωνία επενδυτική, γιατί να πας τραβά τα πράγματα, γιατί χρειάζεστε προστασία. Θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι το επιχειρηματικό μοντέλο για αυτή τη χώρα, πώς μπορείτε να βοηθήσετε την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό θα ήθελα να ξέρω. Ε, βγάζοντας και πάρα πολλά κέρδη. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Η ΣΚΑ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κάποια ερωτήματα προς την Κομισιόν. Πώς βλέπετε τη διάκριση των εθνωτικών κοινοτήτων στην ε, Μιανμάρ και τι θα κάνουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν ξέρουμε για κάτι τέτοιο. Εγώ ανησυχώ. Γιατί, σέντουμε, γιατί στέλνουμε το ίδιο μήνυμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι όλα πάνε καλά. Είχαμε τη συζήτηση στο παρελθόν με τα παραδείγματα των ΗΠΑ κτλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή θέλουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ΗΠΑ και παραμένοντας στο θέμα των ΗΠΑ είπατε ότι θα εφαρμόσουμε πάντα τα ίδια πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Εδώ όμως έχουμε διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι οι ίδιε καταστάσει στι ΗΠΑ και στην Μιανμάρ. Μήπω θεωρεί η Κομισιόν πρέπει να δούμε τα πράγματα στην πραγματικότητα και να έχουμε την, ε, μια συμφωνία που ακολουθεί την πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν περισσότερα προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ό,τι έχουμε στι ΗΠΑ. Ναι, ναι, Και η Συμφωνία Επενδύσεων θα ακολουθήσετε το κλασικό μοντέλο όπως τη συμφωνία με τον Καναδά, παραδείγματος χάρη, ή θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό. Ο κ. Ντάτμουθ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χωρίς να είμαι ε, χωρίς να μην είμαι αυρόφρον, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φερστάπεν για την παρουσίασή του. Μακάρι να ακούγαμε περισσότερους να λέει τέτοια πράγματα. και θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία την κυρία Μάινα η οποία και αυτή ήταν πάρα πολύ εύγλωτη. Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα που έχουμε εδώ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψη των πολιτικών της αριστεράς. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανέφερε ο Ντέβιτ Μάρτιν, ακροθυγός. Τα στοιχεία που έδωσε ο κ. Φεστάπεν και δεν τα κατέγραψα όλα, είναι ότι ο κύριος επενδύστη στη Μιανμάρα αυτή τη στιγμή είναι η Κίνα. 14 δισεκατομμύρια δολάρια είπατε. Σε σύγκριση, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 2 με 200 με 600 εκατομμύρια δολάρια. Και οι επενδύσεις ε, από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ χαμηλή, πολύ χαμηλές. Υπάρχει μια ανησυχία Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν την πολιτικοποίηση του εμπορίου. Αλλά, αλλά εδώ έχουμε ένα χτυπητό παράδειγμα στη Μιανμάρ. Πέρασα από εκεί το 1970 και καταλαβαίνετε τώρα πόσο χρονών είμαι, ενώ φαίνομαι νεότερος. Ήταν σαν μια τροπική ανατολική Γερμανία τότε. Και τα πράγματα μάλλον έχουν βελτιωθεί. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να θέσω ως ερώτημα είναι αν πείτε δεν θα αγγίξουμε τη Μιανμάρ, εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πάμε στη Μιανμάρ και μπορώ να καταλάβω την επιχειρηματολογία την οποία σέβομαι που λέει κάτι τέτοιο. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι άλλες χώρες, στην πραγματικότητα την Κίνα, που δεν νοιάζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθόλου αν νοιάζεστε λοιπόν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν ξέρω ποια είναι η απάντηση, αντιμετωπίζετε το πρόβλημα του να πείτε εμάς μας νοιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, γι' αυτό πιστεύουμε ότι οι εταιρείε της Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να πλησιάσουν τη μα Το αποτέλεσμα είναι ότι όλε οι επενδύσει έρχονται από την Κίνα που σκασίλατσε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τίποτα από ότι εμεί σεβόμαστε βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν πρόκειται να επηρεάσουν τι θα κάνει η Κίνα στη Μιανμάρ. Απλώς θέτω αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής. Ε, θέλω μέσω του Προέδρου να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Θα υποστηρίζετε να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτό που κάνουμε με τα, με τα κράτη που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή να υπάρχει ένα μεταβατικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να προσεγγίσουν το επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θρησκευτική ανεκτικότητας, ελευθερίας λόγου, ένα σύστημα δικαίου, δημιουργία εργατικών ενώσεων κτλ. Και μέχρι ότι όλα αυτά τα πράγματα γίνουν πραγματικότητα μάλλον όταν γίνουν αυτά τα πράγματα τότε χαλαρώνεται τους περιορισμούς και αρχίζεται το εμπόριο με ένα τέτοιο κράτος. Θα το σκεφτόσασταν κάτι τέτοιο για τη Μιανμάρ. Και εγώ να προσθέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν για την συμφωνία επίλυσης διαφορών με τους επενδυτές. Μιλάτε πάντα για τα δικαιώματα των επενδυτών. Μήπως πρέπει να συζητήσουμε και τις υποχρεώσεις των επενδυτών, ιδίως στην ε, περίπτωση της Μιανμάρ. Ποιος θέλει να αρχίσει να δώσει απαντήσεις, ο κ. Πούλμαν. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κ. Φεστόπεν δεν είναι Ολλανδός, αλλά μιλά πολύ καλά. Εγώ είμαι όμως. Yes, and you, you, um, your question starts actually on two sides. Uh, Είχα οι δύο πτυχέ ερώτηση. Πρώτα την κερδοφορία και δεύτερον ε, τι προσδοκίε έχουμε. Έχουμε μακροπρόθεσμη θεώρηση των πραγμάτων των σχέσεων με τη Μιανμάρ. Είναι πολλαπλά τα προβλήματα, δεν περιμένουμε να επιληθούν γρήγορα. και οι πρόκληση που αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε που είναι επιχειρηματικού τύπου και πρέπει να επιλύονται τις επιχειρήσεις είναι δύσκολα προβλήματα και χρειάζονται χρόνο. Οπότε αρχικά όχι, δεν θα έχουμε κέρδη. Σκληρή δουλειά, κατάρτιση, δημιουργία ικανοτήτων, δημιουργία υποστήριξης κλπ. αφορά η πρώτη περίοδος θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων γιατί δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και είναι εμπόδιο για τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Αυτό είναι ο βασικός στόχος αρχικά. Και σαν αποτέλεσμα αυτού τα πρώτα χρόνια δεν περιμένουμε να έχουμε κέρδη. Όμως περιμένουμε να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και την εταιρεία που θέλουμε να δημιουργήσουμε εκεί. Και μακροπρόθεσμα θα έχουμε κέρδη. Αναμένουμε ότι όταν ξεκινάμε σε μια κοινοπραξία με ντόπιο εταίρο, κάτι που προτιμούμε, διότι έτσι λαμβάνουμε υπόψη ντόπιες ευαισθησίες που έτσι ξέρουμε εμείς. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε τη γνώση τους. Προτιμούμε λοιπόν να εργαζόμαστε έτσι σε κοινοπραξία. Και θέλουμε και τα δύο μέρη και εκείνοι να προστατεύονται. Εάν λοιπόν το κάνουμε αυτό και το λάβουμε υπόψη, οι ευρωπαϊκές χώρες, οι ευρωπαϊκές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν πολύ, ε, να βοηθήσουν τις εταιρείες της Μιανμάρ και αντιστρόφως. Και με αυτή την προσέγγιση συνολικά είναι βιώσιμη. Ένα σύντομο σχόλιο παρακαλώ. Πολύ σύντομο. Μισό λεπτό λέει ο Πρόεδρος. Μισό λεπτό. Συνάδελφοι και φιλοξενούμενοι. Τώρα θα συνεχίσουμε στα αγγλικά διότι σταματούν οι διερμηνείς. Σας ευχαριστούμε. Καλή σας όρεξη πλευράς διερμηνέων. Uh, and we stick to English. Mr. Verstappen has very short comment. Thank you for. Belgian, so thank you. <laughs>